Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω θερμά στην απογευματινή μα ακρόαση. Μια και μερικοί εμπειρογνώμονε μας είναι και καθηγητές πανεπιστημίου, τηρούμε τις πανεπιστημιακές παραδόσεις, δηλαδή το τέταρτο το πανεπιστημιακό για την έναρξη το... της ακρόασης. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα πολύ σημαντικό θέμα στη δημόσια ακρόαση. Τους μηχανισμούς για τη μείωση της αστάθειας των τιμών στις γεωργικές αγορές. Είναι σημαντικό αυτό το πρόβλημα και πλήττει ιδιαίτερα τους γεωργούς. Γιατί είναι δύσκολο να ε, έχει κανείς μια γεωργική εκμετάλλευση και να είναι βιώσιμη αν ε, η τιμή για τα προϊόντα του και την εισοδιά του υπόκειται σε τόσο σημαντικές διακυμάνσεις και μάλιστα είναι και απρόβλεπτη. Δύσκολο είναι με τέτοιους όρους να λάβει κανείς και επενδυτικές αποφάσεις. Ως συνήθως έχουμε προσκαλέσει εμπειρογνώμονες για τη δημόσια κρόαση θα μας βοηθήσουν στην ανάλυση του σημαντικού αυτού θέματος και θα μας παρουσιάσουν τις απόψεις τους, τα συμπεράσματά τους, τα πορίσματα που προέκυψαν από τις έρευνές τους, θα μοιραστούν μαζί μας τις εμπειρίες τους. Έχουμε καλεσμένους τους οποίους θα σας παρουσιάσω με τη σειρά που θα μιλήσουν. Ο κύριος Πατρίκ Φερέρ είναι Γενικός Γραμματέας του Επιστημονικού Επιτελείου του Think Tank safagr id Ασχολείται με την ε, με τις ιδέες και την πολιτική για την γεωργία και το... την γεωργική οικονομία. Ο κύριος Φελίτσε Αντινόλφ είναι καθηγητής γεωργικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον κύριο Γερούν επίσης πανεπιστημιακό, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της ε, Γάνδης, που επίσης θα μας μιλήσει για τη γεωργική οικονομία. Κατόπιν θα ακούσουμε τον κύριο Λίαν Φέντον, που είναι διευθύνων σύμβουλος της FC Stone Europe, μιας ε, ιδιωτικής επιχείρησης ε, που παρέχει σε πελάτες ανά τον κόσμο συμβουλές ε, για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και προσπαθεί να τους βοηθήσει να διαχειριστούν καλύτερα αυτή την αστάθεια και τις μεγάλες διακοιμάνσεις των τιμών. Κατόπιν θα μιλήσει ο κύριο Ζακάλ, που είναι Γενικό Γραμματέα ε, του Επιστημονικού Επιτελείου του Think Tank Momagri. Ε, ένα επιτελείο που αναπτύσσει προτάσεις για τη ρύθμιση των γεωργικών αγορών σε παγκόσμια κλίμακα. Θα ήθελα να του ευχαριστήσω όλους θερμά για την ε, έλευσή τους στις Βρυξέλλες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα στην Επιτροπή Γεωργίας και περιμένουμε με ανυπομονησία τα σχόλιά σας, γιατί όπως ξέρετε πρόκειται να εκπονήσουμε και έκθεση πρωτοβουλίας με το θέμα αυτό. Μια έκθεση που θα συντάξει η συνάδελφος Ανζελίκ Ντελαέ. Οπότε η σημερινή δημόσια κρόση είναι ουσιαστικά το εναρκτήριο λάκτισμα της διαδικασίας που θα καταλήξει στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης πρωτοβουλίας. Ως συνήθως έχουμε το πρόβλημα της κατανομής ε, του χρόνου μεταξύ των καλεσμένων μας και των ευρωβουλευτών. Θα σας ε, παρακαλέσω θεμά να τηρήσετε το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Φερέρ, Πατρίκ Φερέρ. Όπως σας είπα, ο χρόνος ε, είναι περιορισμένος, 8 λεπτά, άντε το πολύ εννέα. Αλλά παρακαλώ μην ξεπεράσετε το 9 λεπτό για να προλάβουμε και να μας μείνει χρόνος για ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση κατόπιν. Οπότε θα ήθελα πρώτα να δώσω το λόγο στον κύριο Φερέρ για την εισαγωγή. Επαναλαμβάνω ένα εγκάρδιο καλωσόρισμα προς όλους τους καλεσμένους μας. Κύριε Φερέρ, σας ακούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αστάθεια μπορεί να μετρήσει το μέγεθος και την ταχύτητα της εξέλιξης της τιμής ε, ε, ενός ε, εμπορεύματος σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Στην οικονομική θεωρία, η αστάθεια συνδέεται με δύο έννοιες, ε, την αβεβαιότητα και την μεταβλητότητα. Η μεταβλητότητα των τιμών, δηλαδή οι μεταπτώσεις τους, είναι ένα ε, σύνηθες και κανονικό στοιχείο της λειτουργίας των ε, αγορών. Ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση μεταβάλλεται και η τιμή. Όμως αυτή η κανονικότητα αλλάζει όταν ε, γίνονται αβέβαιες αυτές οι μεταπτώσεις και υπόκειται σε πολύ μεγάλες μεταβολές. Στα γεωργικά ξέρουμε ότι υπάρχει μια ανελαστικότητα της, ε, ε, του λόγου προσφοράς και ζήτησης. Ξέρουμε και τον περίφημο νόμο King. Οι τιμές των γεωργικών προϊόντων πάντα βέβαια είχαν μεγάλες μεταπτώσεις, όμως παραδόξως λίγες ε, περιόδους αστάθειας τιμών. Η γεωργική πολιτική, μάλιστα, κατάφερε στο παρελθόν να προστατεύσει τους παραγωγούς από, αυτή την αστάθεια με την υιοθέτηση διαφόρων ε, μέτρων προστατευτικών που από το 1992 όμως έχουν αμφισβητηθεί ε, και ανακληθεί μέσω διαφόρων εξελίξεων και, μετα, και μεταρρυθμίσεων. Όμω βλέπουμε με την αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση των συναλλαγών, με την εξέλιξη ότι αφορά τη γεωργική πολιτική σε Ευρώπη και Αμερική ε, που καταργούν οποιαδήποτε παρέμβαση μέσω αποθήκευση, με την ε, υιοθέτηση χαρακτηριστικών χρηματαγοράς ε, των γεωργικών αγορών, με τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, χωρίς να ξεχνούμε και τις πολιτικές ορισμένων σημαντικών φορέων. Γίνεται λοιπόν η παγκόσμια αγορά πλέον πιο ευαίσθητοι και ευάλωτοι ε, σε τέτοιες περιόδους αστάθειας που είναι πιο ακραίες και πιο συχνές. Ε, επί παραδείγματι, ε, μετά τα φαινόμενα ξηρασίας, μετά την πτώση 2,3% της παγκόσμιας συγκομιδής, όλα αυτά συνδυασμό και με το εμπάργκο με τις εξαγωγές στη Ρωσία ή ε, αγορές ε, υπεραντιδρούν με μία αύξηση κατά 70% ε, των τιμών στα άλευρα, στα σιτηρά. Βλέπουμε ότι σήμερα επιμένουμε πιο πολύ σε πολύ σημαντικές μεταπτώσεις, ημερήσεις ή εβδομαδιαίες μεταπτώσεις που παλαιότερα τις παρατηρούσαμε σε μια περίοδο ετήσια για παράδειγμα. Και οι κλιματικές αλλαγές δεν είναι και αυτές ε, προβλέψιμες. Γι' αυτό το λόγο έχουμε θέσει συγκεκριμένα αποθέματα αποθήκευσης για να έχουμε ε, μία στρόφιγγα αν θέλετε την οποία μπορούμε να ανοίγουμε ή να κλείνουμε ανάλογα με, το πλεόνασμα ή την έλλειψη συγκεκριμένων προϊόντων. Ε, μάλιστα οι τιμές αυξήθηκαν ε, πάρα πολύ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και μάλιστα αυτό οδήγησε σε υπερπαραγωγή. Όμως ούτε αυτό είναι λύση. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η υιοθέτηση χαρακτηριστικών χρηματαγοράς στα γεωργικά προϊόντα έχει εντείνει την αστάθεια. Σε περίοδους κρίσης οι όγκοι ε, που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών ε, τετραπλασιάζονται ή και οκταπλασιάζονται. Και εδώ η πλαισίωση σε ό,τι αφορά τις ε, πιστώσεις ε, και τις δεσμεύσεις ε, πληρωμών είναι κάτι που προβάλλεται ως λύση, όμως και εδώ η κερδοσκοπία μας επηρεάζει. Όπως και να έχει, υπάρχει μία γενική αναγνώριση των αρνητικών προεκτάσεων της ευρύτερης αστάθειας των τιμών, που διακινδυνεύει τα έσοδα και το μέλλον των παραγωγών. Από την άλλη και οι πολύ ψηλέ ε, τιμέ ε, ουσιαστικά τιμωρούν τις χώρες που δεν έχουν επιστημική ασφάλεια και είναι και συνήθω οι πιο φτωχές χώρες. Και έχουμε μιλήσει και ε, για διάφορες αναταραχές που έχουν προκύψει ως απόρρια της πείνας. Είναι αρκετά η κατάσταση. Γι' αυτό και το 2011 ε, το G20 στο Παρίσι εξέτασε ένα σχέδιο δράσεων για να καταπολεμήσουμε αυτή την αστάθεια. Να επενθυμίσουμε τα πιο κύρια σημεία. Να αυξήσουμε την παραγωγή και τη γεωργική παραγωγικότητα. Διεθνής ε, πρωτοβουλία για την έρευνα για την βελτίωση των σιτήρων. Το πρόγραμμα ERV. Δεύτερον, να βελτιώσουμε την ενημέρωση διαφάνεια των αγορών. Το σύστημα AMIS του για την ε, αναγνώριση των αποθεμάτων και η Διεθνής Πρωτοβουλία GeoGlam ε, για να εξετάσουμε και τι συμβαίνει με την ε, δορυφορική παρατήρηση καθώς και ένα φόρουμ άμεσης ανταπόκρισης και απαγόρευση του περιορισμού ή της φερολόγησης για την επιστημιστική βοήθεια του Παγκοσμίου προγράμματος ε, του επιστηστικού. Μετά, το ΙΟΣΚΟ έχει επιφορτιστεί ε, την ε, ρύθμιση των χρηματαγορών σε ό,τι αφορά τις αγορές παραγόγων πρώτων υλών. Τώρα, ορισμένε παρατηρήσει. Το G20 συνήλθε το 2011 και δεν έχουν υπάρξει σημαντικέ εξελίξει ό,τι αφορά το σχέδιο δράσεων. Η η υπερβολική αστάθεια συνεχίζει και προς τις δύο μεριές μάλιστα. Ορισμένες χώρες θεωρούν ότι τα επίπεδα αποθεμάτων τους είναι στρατηγικά δεδομένα και έτσι εμπιστευτικά διαπραγματισμένα και έτσι δεν τα μοιράζονται με άλλους. Ε, σε ό,τι αφορά την πλαισίωση της παραγωγής είναι κάτι το ενδιαφέρον, όμως σε διεθνές επίπεδο ε, συμφέρει περισσότερο και ενδιαφέρει αυτούς που δεν τα εφαρμόζουν στην πράξη. Η κρίση του 2008-2009 μας οδήγησε τελικά σε μεγάλη ρευστότητα στην αγορά και έτσι προέκυψε ο πειρασμός ε, ορισμένων που ε, ενέδωσαν και έτσι έδωσαν μεγαλύτερο έναυσμα σε αυτή την αστάθεια. Έχουν περάσει περίπου τέσσερι δεκαετίες με προστατευμένε αγορές, με ε, εγγυημένες τιμέ. και τώρα βλέπουμε ότι η γεωργική πολιτική παραμένει ανοιχτή ε, στον υπόλοιπο κόσμο. Η αστάθεια έχει μπει στι αγορές μας ε, και στου κλάδους μας και οι κλάδοι μας υφίστανται τι συνέπειε, ιδίω σε παραγωγή. Περιμένουμε μία ευωτιθέμενη διεθνή ανταπόκριση στην κατάσταση, όμως πρέπει να αντιδράσουμε πραγματικά, ούτω ώστε κάθε επεισόδιο τέτοια αστάδειας να μην μεταφράζεται σε μία περίοδο αναδιάρθρωσης για τη γεωργική πολιτική στα κράτη-μέλη. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Φερέρ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Σαντινόλφη που θα μας μιλήσει για τους υπάρχοντες ε, μηχανισμούς ε, για την αντιμετώπιση της αστάθειας των τιμών, ιδιαίτερα στην κοινή γεωργική πολιτική. Δικαιούστε και εσείς ένα οκτάλεπτο κύριε Αντινόλφη, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ και τους συναδέλφους από το Τμήμα Πολιτικών. Εγώ θα ήθελα στην ε, ομιλία μου να ξεκινήσω. Παρακαλώ, ας περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ βλέπετε μια σύνοψη της παρουσίασής μου. Φυσικά ε, λίγο είναι ο χρόνος. Θα προσπαθήσω να σας μιλήσω για τα αίτια της αστάθειας των τιμών, τους παράγοντες που επηρεάζουν ε, ε, το εισόδημα το γεωργικό και τους, κινδύνου κινδύνους που υπάρχουν γι' αυτό Επίσης ε, θα σας παρουσιάσω τους μηχανισμούς που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της στάθειας των τιμών και την διαχείριση των κινδύνων. Θα σας παρουσιάσω και τα παραδείγματα του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών και τα δικά τους νομοθετικά πλαίσια και στο τέλος θα υποβάλω και κάποιες συστάσεις, κάποιες προτάσεις ε, για τη μελλοντική μεταρρυθμίση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Έχω κάποια προβλήματα με τις διαφάνειες και τη σειρά δυστυχώς που εμφανίζονται, αλλά θα τα καταφέρω πιστεύω. Όπως είπε και ο συνάδελφος, η αστάθεια των τιμών ε, συνδυάζεται άμεσα με βασικούς παράγοντες αγοράς, την προσφορά και τη ζήτηση. Τα τελευταία χρόνια προστάθηκαν και, άλλοι, και άλλες μεταβλητές μακροοικονομικού χαρακτήρα πολύ σημαντικοί κυρίως όσον αφορά τις ε, σχέσεις ανάμεσα στα γεωργικά προϊόντα και άλλα προϊόντα. Όσον αφορά το θέμα των αποθεμάτων, ε, το θέμα της εμπορικής ε, πολιτικής, όλα αυτά είναι ένα θέμα το οποίο σε μεγάλο βαθμό βρίσκεται σε αντίδραση και σε αναντιστοιχεία με τις άλλες αγορές. Βλέπετε λοιπόν ότι την περίοδο 7, 8 και κατά την περίοδο 10-11 υπάρχει μια περιπλοκότητα όσον αφορά τους οικονομικούς παράγοντες. Είναι ένα πολύ περίπλοκο φαινόμενο και σε αυτό συμβάλλουν διάφορα στοιχεία. Όπως βλέπουμε εδώ υπάρχουν παράγοντες αντίξωοι, ε, κλιματικοί, εμπορικοί, το επίπεδο των αποθεμάτων, ε, η υποτίμηση του δολαρίου. Είναι μία σειρά θεμάτων τα οποία τροφοδοτούν αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ε, αστάθεια τιμών Όλα αυτά έχουν ε, αναζωογονήσει τη συζήτηση για το όλο θέμα και προβάλλονται περισσότερο και από τα μέσα ενημέρωσης. Η αστάθεια λοιπόν των τιμών επηρεάζει αρνητικά τον γεωργικό τομέα. Στην ε, περίπτωση της Ευρώπης ε, πέρα από τα παραδοσιακά προβλήματα που έχουν σχέση με την ατέλεια των μηχανισμών ε, των τιμών ε, στις αγορές ε, και σε συνδυασμό με χρηματοοικονομικά προβλήματα που έχουν σχέση με την γεωργική πολιτική. Πέρα από όλα αυτά έχουμε και μια πολύ σημαντική θεσμική αλλαγή. Σε αυτό αναφέρθηκε και ο συνάδελφος. Τα τελευταία 25 χρόνια έχει προκύψει, έχουν προκύψει σημαντικές αλλαγές, κυρίως αν δούμε το θέμα της αστάθειας των τιμών και της διαχείρισης των κινδύνων. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περιορίσει την προστασία των γεωργών και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστική αναθεώρηση ε, του, του, του τρόπου με τον οποίο μπορεί κανείς να στηρίξει το αγροτικό εισόδημα. Όσον αφορά λοιπόν αυτά τα θέματα, δεν ξέρω πού πρέπει να σημαδεύω για να το ρυθμίσω τον υπολογιστή. Έχω κάποια, κάποιο τεχνικής φύσεως πρόβλημα, δεν ξέρω τι να κάνω, λέει ο μιλητής. Τέλος πάντων, ε, όσον αφορά λοιπόν ε, αυτά τα θέματα της διαχείρισης κινδύνων στην ε, δική μας την παρουσίαση αναφέρουμε τρεις περιπτώσεις της Ευρώπης που γνωρίζουμε πολύ καλά, όπου έχουμε από τη μια ε, τις αγορές και από την άλλη τις ενισχύσεις προς τους ε, γεωργούς. Κατόπιν έχουμε όλα τα μέτρα του δεύτερου πυλώνα που κατ' ουσίαν περιλαμβάνουν τις ε, στρατηγικές ε, που μπορούν να εφαρμοστούν εκ των προτέρων για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που απορρέουν από αντίξωες συνθήκες. Και κατόπιν έχουμε αυτό που λέμε ε, Risk Management Toolkit, δηλαδή προστασία εναντί των φυσικών καταστροφών σε περίπτωση που προκύψουν κάποιες επιδημίες ε, ή φυσικές καταστροφές. Το τρίτο αυτό στοιχείο είναι πολύ σημαντικό και είναι και μια καινοτομία σε σχέση με αυτά που προσφέρονται ε, στους ε, γεωργούς. Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να υπάρχει ένα ταμείο αμοιβεοποίησης το οποίο να καλύπτει κινδύνους για το εισόδημα των γεωργών. Δηλαδή θα μπορούσαν να υπάρξουν ε, σημαντικές μειώσεις του εισοδήματος και αυτό το εργαλείο το οποίο σε τελική ανάλυση βρίσκεται σε πειραματική φάση σε κάποιες χώρες, στην Ιταλία, στο Βέλγιο, στη Φλάνδρα. Αυτό ε, ενδιαφέρει ιδιαίτερα διότι κατ' ουσίαν είναι το μόνο εργαλείο το οποίο επιτρέπει κατά κάποιον τρόπο να διαχειριστούμε τους κινδύνους επί των τιμών. Κατόπιν προσπαθήσαμε να ανοίξουμε και ένα παράθυρο ε, σε σχέση με τον Καναδά όπου ο Καναδάς έχει μία μακρά ιστορία, σε αυτή την εμπειρία της διαχείρισης των κινδύνων. Έχει ένα οπλοστάσιο μέτρων ε, σε σχέση με τους γεωργούς του Καναδά. Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο, γιατί κατά κάποιον τρόπο είναι καινοτόμο, είναι το τι μπορούμε να επιλέξουμε ως βάση αναφοράς και αναφέρομαι στο σύστημα AgriDisk, το οποίο δεν εφαρμόζεται ευρέως, όμως ε, το μοντέλο αυτό επιτρέπει ε, κατά κάποιον τρόπο AgriRisk να έχουμε έρευνα σχετικά με το μοντέλο που σας είπα, το AgriRisk, ε, δηλαδή το πώς μπορεί κανείς να χειριστεί την το πρόβλημα αυτό. Αυτό λειτουργεί κατ' ουσίαν μέσω ενό λογαριασμού. Δηλαδή για κάθε, για κάθε γεωργό υπάρχει ένας λογαριασμός όπου γίνεται συγχρηματοδότηση και από το κράτος. 1% είναι το ποσοστό που χορηγείται από το κράτος και αυτό βοηθάει τους γεωργούς ε, σε περίπτωση που έχουν ε, ζημιές, απώλειες. Όταν έχουν προβλήματα μπορούν να τρέξουν εκεί για να έχουν ένα κεφάλαιο κίνησης. Και έτσι λοιπόν οι γεωργοί μπορούν να έχουν κάποια σιγουριά, να νιώθουν κάποια ασφάλεια, ε, ότι θα αντιμετωπίσουν κινδύνους και μπορούν να κάνουν και μακρόπνοες επενδύσεις το ε, Stability είναι εκείνο που μοιάζει περισσότερο με το δικό μας το, σύστημα είναι κατ' ουσίον μία παρέμβαση της κυβέρνησης τη στιγμή που υπάρχουν ε, ζημιές πάνω από 70% σε σχέση με τη βάση αναφοράς όπου ε, στην, στον Καναδά είναι ένα δολάριο για κάθε χίλια διασφαλισμένα ευρώ. Ας δούμε λιγάκι την εμπειρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν θα αναφερθώ διεξοδικά σε αυτό. Ε, υπάρχει μία μελέτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που συγκρίνει το τι συμβαίνει στι ΗΠΑ και τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Και εκεί υπάρχουν πάρα πολλέ ενδιαφέρουσε λεπτομέρειε. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να δούμε ότι με το τελευταίο νόμο σχέδιο που θεσπίστηκε στι ΗΠΑ ολοκληρώθηκε μία διαδικασία η οποία προβλέπει την πλήρη κατάργηση των άμεσων πληρωμών. Αυτά υποκαθίστονται με συστήματα διαχείρισης κινδύνου. Δηλαδή διάφορα προγράμματα τα οποία ε, εμφαρμόζονται παράλληλα με ε, πληρωμές που είναι αντικυκλικές και όχι άμεσες. Βλέπουμε λοιπόν ε, το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, το βλέπετε στο γράφημα. Εκεί βλέπουμε την, ε, τον επιμερισμό των πόρων σε δύο χώρες και οι διαφορές είναι έντονες. Υπάρχει πολύ σημαντικό ανώτατο όριο, αυτό το διαπιστώνουμε τα τελευταία χρόνια και Όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων, ε, μπορείτε να δείτε στο γράφημα την κατάσταση που υπάρχει στην Ευρώπη, όπως επίσης ε, και την στήριξη των εισοδημάτων. Στις ε, Ηνωμένε Πολιτείε είναι η μικρότερη στήριξη από ό,τι στην Ευρώπη. 30 δευτερόλεπτα μου μένουν ακόμα. Έχασα χρόνο με αυτές τις τεχνικές τέλος πάντων δυσκολίες που έχω. Βλέπουμε όμως ότι στο μέλλον θα μπορούσαν να υπάρξουν πολλές ευκαιρίες να ξεκινήσουμε από αυτή την ε, καινοτομία έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα σύστημα το οποίο θα είναι πιο ευέλικτο, το οποίο θα μπορεί κατά κάποιον τρόπο τις άμεσες πληρωμές να τις ε, αναδιαμορφώνει όχι μόνο κάτω από το πρίσμα το χρηματοοικονομικό αλλά και από το πρίσμα του ότι η Ευρώπη μπορεί να, κάνει, να καταβάλει περισσότερες ε, προσπάθειες όσον αφορά στη γεωργία. Στη Γαλλία ε, λειτουργήσε αυτό το σύστημα και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πλαίσιο έτσι ώστε εκεί να μπορούν να συμμετέχουν με μονομένη γεωργία έτσι ώστε να είναι δυνατόν σε περίπτωση ζημιάς να μπορεί κανείς να παρέμβει αλλά όταν η ζημιά είναι πολύ μεγαλύτερη τότε είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, κάποια αντιστοιχεία με τον προβολισμό. Ξεπέρασα κατά το χρόνο μου, ζητώ συγγνώμη και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντινόλφη. Το λόγο έχει τώρα ο καθηγητής Μπούισε από το Πανεπιστήμιο της Γάνδης. Παρακαλώ. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να σας δώσω πρώτα κάποιες διεξοδικές εξηγήσεις για αυτά που ακούσαμε πριν από λίγο από τον συνάδελφο, γιατί υπάρχει διαφορά μεταξύ της ευρωπαϊκής πολιτικής και της πολιτικής των ΗΠΑ, γιατί η δική μας πολιτική στον πυλώνα 1 δίνει στήριξη εισοδήματος άσχετα με την κατάσταση των αγορών. Ο συνάδελφος μας το ανέφερε ως ε, ε, θέμα ε, εισοδήματος και όχι διαχείρισης κινδύνου. Μερικοί θα το θεωρούσαν ως ε, μηχανισμό διαχείρισης κινδύνου, γιατί λαμβάνουν οι γεωργοί κάποιο ποσό. Στι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν μακρά ιστορία ε, τέτοια αντικυκλική στήριξη του τομέα. Είναι σημαντική λοιπόν αυτή η διαφορά των δύο συστημάτων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτείων και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη, επίσης στις σε εμά έχουμε το, το πυλώνα 2 και τη στήριξη του εισοδήματο και κάποιες άλλες πολιτικές προαιρετικές στον πυλώνα 2 που δεν εφαρμόζουν όλες ε, οι χώρες μέλη, δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε ένα πρόγραμμα προστασίας του περιθωρίου στο γαλακτοκομικό τομέα με ομοιόμορφη εφαρμογή. Επίσης υπάρχουν ε, ε, συστήματα για την προστασία του περιθωρίου και στα θέματα των ε, ζωοτροφών, αλλά έχουν καθεστώτα που ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες του κάθε γεωργού. Εμείς έχουμε ε, την ασφαλιστική δικλίδα τη βοήθεια για την ιδιωτική αποθεματοποίηση, που είναι ελάχιστη συμβολή στο θέμα τη διαχείριση του κινδύνου από πλευρά Γιώργου, αλλά παρόλα αυτά κάπω βοηθάει. Υπάρχουν πολιτικέ πρόθεσεις, υπάρχουν άμεσε πολιτικέ που συμβάλλουν άμεσα στη διαχείριση του κινδύνου για του γεωργού. Επίση, ε, έχουμε και τι οργανώσει παραγωγών που με τα επιχειρησιακά του προγράμματα μπορούν να κάνουν απόσυρση προϊόντων από την αγορά. Α μην το ξεχνούμε και αυτό είναι μηχανισμός διαχείρισης κινδύνου. Και για να συνεχίσω αυτά που είπα προλαλή σας, ε, θα ήθελα να πω ότι για τις γεωρικές πολιτικές ε, να δούμε και τις άλλες αγορές ε, σε άλλα προϊόντα και άλλες υπηρεσίες πώς αντιμετωπίζουν την αστάθεια των τιμών. Για παράδειγμα, αγορά ηλεκτρικού ρεύματος είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος, όπως στα τρόφιμα, θέλουμε ένα σταθερό ανεφοδιασμό. Και επίσης έχουμε απελευθερωμένη αγορά στην αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρικής ενέργειας. Εκεί ε, υπάρχει ελεύθερη απόφαση για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν επίσης αγορές ε, ε, προθεσμιακές, μακροπρόθεσμες στην ηλεκτρική ενέργεια. Το ίδιο ισχύει και για τις αγορές τροφίμων. Υπάρχουν αυτές οι προθεσμιακές συμβάσεις. Επίσης, στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, οι θύνοντες της πολιτικής αναγνωρίζουν την ανάγκη παρέμβασης, προκειμένου η αστάθεια των τιμών να μην αντιμετωπιστεί μόνο από τις προθεσμιακές ε, αγορές, τις future markets, αλλά όχι μόνο από την παραγωγή, αλλά και τη δυνατότητα παραγωγής, γιατί σε περισσότερες χώρες υπάρχει ε, ένα, ένα δυναμικό παραγωγής και δίνεται ε, στήριξη είτε για, για κλείσιμο, είτε για αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπου χρειάζεται. Κάτι τέτοιο ανταποκρίνεται και στις ευρωπαϊκές πολιτικές με τη μορφή που έχουν σήμερα, γιατί οι γεωργοί λαμβάνουν στήριξη του εισοδήματο. Για να το πετύχουν όμως θα πρέπει να κρατήσουν την γεωργική γη, τα γεωργικά εδάφη σε καλές, σε καλές συνθήκες καλλιέργειας. Στο παρελθόν η υποχρέωση αγρανάπαυση ήταν κάτι αντίστοιχο στην κοινή γεωργική πολιτική, θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά δεν υπάρχει σύστημα που όταν έχουμε υπερβολική προσφορά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τι ε, ενισχύσει για να μειώσουμε την προσφορά και να αντιμετωπίσουμε την πλεονασματική προσφορά σε κάποιο προϊόν. Γιατί κάτι τέτοιο υπάρχει στην ε, αγορά ηλεκτρική ενέργεια, αλλά δεν υπάρχει στην αγορά τροφίμων. Κάποια χαρακτηριστικά είναι κοινά και στι δύο αγορές, τη γεωργικής ε, παραγωγή και τη παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια. Οπότε θα μπορούσαμε ίσω να διδαχθούμε από την αγορά ηλεκτρική ενέργεια για τη μελλοντική μα διαχείριση. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν θα πρέπει να κλείνουμε τι αγορέ ω λύση για να λύσουμε την αστάθεια των τιμών. Δεν είναι αυτή η λύση ούτε και για την ηλεκτρική ενέργεια. Άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι η διαφάνεια και η ενημέρωση θα πρέπει να είναι προσιτέ σε όλου του παράγοντε αγορά. Είναι σημαντικό και για την ηλεκτρική ενέργεια αλλά και για την αγορά γεωργικών προϊόντων. Δεν θα πρέπει να στηρίζουμε την παραγωγή όταν υπάρχει ε, υπερβολική προσφορά. Στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας σε μερικά κράτη-μέλη έχουμε ενίσχυση για ηλεκτρισμό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, άσχετα με το σημείο ε, τη στιγμή παραγωγή τη ενέργεια. Αυτό όμω οδήγησε σε αρνητικές τιμέ του ηλεκτρισμού, του ηλεκτρικού ρεύματο. Είχαμε δηλαδή παραγωγή ε, ηλεκτρική ενέργεια όταν το ε, δίκτυο ήταν ήδη πλήρες θα πρέπει στη γεωργική πολιτική να δίνουμε κίνητρα για αύξηση της παραγωγής, όχι όμως όταν υπάρχει ήδη η πλεονασματική προσφορά στην αγορά. Κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε ως ιδέα είναι να δούμε πώς ε, θα ενισχύσουμε το δυναμικό και όχι την παραγωγή. Και όταν υπάρχει πλεονασματικό δυναμικό να χρησιμοποιήσουμε τις επιδοτήσεις για να χρησιμοποιήσουν λιγότερο μεταβλητές εισρωές οι Γεωργή. Γιατί σήμερα έχουμε μεγάλα αποθέματα στις αγορές ετηρών. Τι θα κάνουμε όμως αυτή την άνοιξη. Οι ε, γεωργοί θα χρησιμοποιήσουν ε, όσο δυνατό περισσότερα λιπάσματα και αζωτούχα κυρίως για να αυξήσουν την παραγωγή. Το θέμα είναι να χρησιμοποιήσουμε τις επιδοτήσεις για να μειώσουμε τον αριθμό των λιπασμάτων και μάλιστα προαιρετικά. Έτσι να αντιμετωπίσουμε το διαφυγό κέρδος από τη λιγότερη προσφορά. Και έτσι θα επηρεάσουμε την σταθερότητα των τιμών και θα κάνουμε και κάτι καλό για το περιβάλλον με τη μείωση της χρήσης των λοιπασμάτων. Αυτά αναλύουμε στο επιστημονικό μας και ερευνητικό μας επιτελείο στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης. Και αυτή είναι και η δική μου συμβολή στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Θα ακούσουμε κάποια σχόλια τώρα. Τα σχόλια θα τα κάνουν πρώτα οι άλλοι καλεσμένοι μας εμπειρογνώμονες. Ο κύριος Καρλ, ένα σύντομο σχόλιο. Δύο-τριών λεπτών. Παρακαλώ κύριε Καρλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, μερικά λεπτά μόνο. Θα ήθελα να πω ότι η διαπίστωση που έγινε από, τους κυρίους, ε, από τον κύριο Φερέρι είναι πολύ σωστή, ότι η αστάθεια τιμών είναι πολύ πιο συχνή, με μεγαλύτερο εύρος ε, μεταβολής των τιμών και η ευρωπαϊκή πολιτική δεν έχει προσαρμοστεί σε αυτήν την κατάσταση. Η μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής δεν μας επιτρέπει πλέον να αντιμετωπίσουμε αυτή την αστάθεια. Δεύτερον, σε διεθνές επίπεδο, οι διαπραγματεύσεις που έγιναν στο πλαίσιο του G20 οδήγησαν σε ένα πρώτο βήμα συνεργασίας ε, σε διεθνές επίπεδο, όμως αυτό είναι ιδιαίτερα ανεπαρκές και όπως ανέφερε και ο κύριος Φερέρ, τα δημόσια αποθεματικά θεωρούνται στρατηγικά και έτσι εμπιστευτικά. Δεν υπάρχει λοιπόν πραγματική διεθνή συνεργασία για τη ρύθμιση των αγορών ή τουλάχιστον για να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις, γιατί η ρύθμιση κατά τη γνώμη μας είναι αυτό, η διαχείριση των κρίσεων που αποτελούν απόρρια τη ε, στάθεια τιμών αυτέ οι κρίσει. Και έτσι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Ο κύριο Οδυνόλφη ανέφερε πολύ σύντομα και την Αμερικανική και Καναδική πολιτική και είπε ότι υπάρχει ένα μέτρο σταθεροποίηση ε, των ε, εισοδημάτων, το άρθρο 39. Το επισημαίνω γιατί αυτό μας επιτρέπει να παρεμβαίνουμε όταν υπάρχει πτώση του εισοδήματο κατά 30%. Φανταστείτε να παρεμβαίνουμε στα, στην αγορά μόνο όταν η πτώση του συστήματος είναι 30%. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι κατάλληλο σαν ε, προσέγγιση. Στον Καναδά έχουμε ένα σύστημα ανάλογα με την προσφορά και ζήτηση και έτσι περιορίζουμε και τις αγωγές. Έχει εξελιχθεί προς ένα σύστημα διαχείρισης κινδύνων και στις ΗΠΑ Πολιτείες. Υπενθυμίζω ότι είναι ένα αντικυκλικό σύστημα που από ε, επιτρέπει τη σταθεροποίηση του εισοδήματο από τη μια χρονιά στην άλλη. Ένα παράδειγμα. Όταν συγκρίνουμε τις ε, παρεμβάσεις των μεγάλων γεωργικών παραγωγών, το 61% στην Ευρώπη είναι ε, αποσυνδεμένες ενισχύσεις που δεν μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, τις κρίσεις, ενώ ας πούμε στις ΗΠΑ, Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία είναι 0% αυτές οι ενισχύσεις. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε αυτό και στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της αστάθειας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Περνάμε στην συζήτηση τώρα. Θα έχουν την ευκαιρία ευρωβουλευτέ να κάνουν τις παρατηρήσεις να υποβάλουν ερωτήσεις. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, παράληψή μου. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Φέντον για ένα σύντομο σχόλιο. Συγγνώμη κύριε Φέντον. Σας ακούμε για ένα σύντομο σχόλιο. Κανένα πρόβλημα. Ένα από του παράγοντε που αναφέρθησαν σε σχέση με την αστάθεια και το κόστος ε, που συνδέεται με αυτήν την αστάθεια και στο πλαίσιο της πράσινης οικονομίας, η πράσινης αγοράς, το βλέπουμε διεθνώς ότι υπάρχουν πολλοί κερδοσκόποι που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις αγορές πολλές ε, έρευνες του ακαδημικού χώρου βλέπουν και καταδεικνύουν που ακριβώς έχει αυξηθεί και που έχει περιοριστεί αυτή η αστάθεια και βλέπουμε ότι είναι μοιρασμένα τα συμπεράσματα. Σε σχέση με την αγορά γαλακτοκομικών εδώ στην Ευρώπη που θα αναφέρω στη συνέχεια και στις διαφάνειές μου ε, βλέπουμε ότι υπάρχει η αστάθεια αλλά δεν έχουμε κερδοσκοπία σε τέτοιο βαθμό σε αυτές τις αγορές. Επομένως, ε, δεν ισχύει απαραίτητο ότι τα ε, χρηματοοικονομικά παράγωγα είναι αυτά που προκαλούν την αστάθεια. Βεβαίως, εγώ εκπροσωπώ τα συμφέροντα της βιομηχανίας και σας το λέω, αλλά θα έλεγα ότι είναι το αντίθετο. Και επίση συμφωνώ με κάτι που αναφέρθηκε ότι χρειαζόμαστε σαφή και ξεκάθαρα διαφανή δεδομένα. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Νομίζουμε ότι θα επωφελήσει τους πάντες γιατί και εγώ σε αγροτική οικογένεια μεγάλωσα και ο αδερφός μου συνεχίζει να εργάζεται σε γεωργική εκμετάλλευση και βλέπω πόσο ε, δύσκολο είναι να λειτουργήσει κανείς μέσα σε έναν κικαιώνα διαφορετικών και αντικρώμενων πληροφοριών ε, και δεν ξέρει τι να ε, πρωτοδιαλέξει. Κάποιοι του λένε ότι θα ανέβει ο τομέα των ενώ είναι σαφές ότι θα πέσει. Επομένω και οι γεωργοί και όσοι συμμετέχουν στην ε, αλυσίδα εφοδιασμού θα μπορούν να παίρνουν καλύτερε αποφάσει σε σχέση με το αν θα πρέπει να αυξήσουν ή να περιορίσουν την παραγωγή του. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Και τώρα περνάμε όντω στη συζήτηση. Πρώτος έχει, ζήτησε το λόγο ο κύριος Ταραμπέλα, παρακαλώ. Ε, έγινε η διαπίστωση και μας την υπενθύμησε και η πραγματικότητα εδώ και κάποια χρόνια. Υπάρχει αστάθεια και μεταβλητότητα πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είχαμε συνηθίσει όταν είχαμε τους μηχανισμούς ρύθμισης. Γιατί αφήσαμε τις ε, συνδεδεμένες ενισχύσεις, δεν έχουμε πια συνδεδεμένες ε, και πάνω από 60% των ενισχύσεων είναι αποσυνδεδεμένες, ενώ οι υπόλοιποι ανταγωνιστές μας διεθνώς ε, εξακολουθούν να, συνδέουν τις ενισχύσεις τους. Επίσης εγκαταλείψαμε τους μηχανισμούς ρύθμισης ε, ε, της προσφοράς στο γάλα, του χρόνου στη ζάχαρη, οπότε αυξάνεται η παραγωγική μας ικανότητα, ενώ η κατανάλωση δεν παρακολουθεί αυτή την αύξηση της προσφοράς και η ζήτηση μένει πίσω. Με, αποτέλεσμα να μειώνονται διεθνώ οι τιμές. Τώρα, τι να πούμε για τι διεθνεί συμφωνίε που είτε έχουμε υπογράψει είτε ετοιμάζουμε και που θα μα οδηγήσουν σε αυξήσει ε, τροφίμων ε, που θα ανταγωνίζονται τα δικά μας, ε, που ήδη παρουσιάζουν υπερπροσφορά. Οποιαδήποτε διεθνή πίεση συμπιέζει τις τιμές προς τα κάτω. Είχαμε πρόσφατα μείωση το τιμών του γάλακτος, ακριβώς επειδή ειχαμε δει είναι δεκατό επιπλέον ποσότητα γάλακτο στις παγκόσμιες αγορές. Ε, βέβαια δεν ξέρω αν αυτό θα πρέπει να το αποδεχτούμε μυρολατρικά ή να προτείνουμε κάποιες λύσεις για να καταπολεμήσουμε αυτή την κατάσταση, γιατί η υπερβολική αστάθεια είναι από τους σημαντικότερους εχθρούς ε, ε, των γεωργών και κυρίως των νέων γεωργών που θέλουν είτε να εισέλθουν είτε να επενδύσουν στο γεωργικό επάγγελμα. Πώς θα καταπολεμήσουμε την υπερβολική αυτή αστάθεια, υπάρχουν μηχανισμοί για να μας βοηθήσουν να το κάνουμε και αν ποιοι είναι οι προτιμότεροι. Επαναφορά των ρυθμιστικών μηχανισμών, ασφάλιση κινδύνων μέσω των ασφαλίσεων, καλύτερη πλαισίωση. Υπάρχουν προτάσεις, ε, έχετε σκεφτεί κάποιες λύσεις. Ευχαριστώ κύριε Referate. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις εισηγήσει που ακούσαμε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα σε αυτά που μας είπε ο καθηγητής από τη Γάνδη. Επιτέλους κάτι ακούσαμε και εδώ ε, σε αυτό το κοινοβούλιο που αναφέρθηκε στον περιορισμό των ποσοτήτων για τη σταθεροποίηση των ε, τιμών. Ακούσαμε κάτι για, τον, για τη διαχείριση των ποσοτήτων του όγκου το να υπάρχει περιορισμός τον όγκο, αυτό έχει επιπτώσει στο σύνολο της αγοράς. Και στην Επιτροπή Γεωργίας ε, λέμε συνέχεια ότι θα πρέπει ίσως ε, να στηρίξουμε την ε, προαιρετική παρέτηση από παραγωγή, ας πούμε, στο γάλα. Αυτό θα μπορούσε, λέμε, να έχει και θετικές συνέπειες για τον Γιώργο γιατί θα χρησιμοποιεί λιγότερες ζωοτροφές και επειδή η αγορά θα έχει λιγότερες διακυμάνσεις θα ωφεληθεί και ο ίδιος. Ακούμε τέτοιου είδους πράγματα. Πάντως ε, αυτή η ομιλία που ακούσαμε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και αυτά που είπαν και άλλοι πολύ ενδιαφέροντα. Ε, κράτησα πολλές σημειώσεις αλλά αυτό που ακούσαμε για την διαχείριση του όγκου αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα χαιρόμουν πάρα πολύ στην Επιτροπή Γεωργίας να συνεχίσουμε τη συζήτηση επί του θέματος αυτού. Διαχείριση του όγκου παραγωγής. Ναι. Θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις ποσότητες. Ο κύριος Ροπέ. Κύριε Ροπέ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι το θέμα της ε, απογευματινής συζήτησης ε, είναι και πολύ σημαντικό και πολύ επίκαιρο. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που μας απασχολεί αυτό το θέμα. Το έχουμε ήδη συζητήσει επανειλημμένως και νιώθω και κάπως αμήχανα και είμαι και σε δύσκολη θέση, γιατί οι προτάσεις που ακούσαμε μέχρι στιγμής δεν είναι και ιδιαίτερα καινοτόμες. Μας μιλήσατε για τις συνέπειες και τα αποτελέσματα, αλλά πού είναι οι προτάσεις για το πώς θα αντιμετωπίσουμε και θα, πώς θα αποτρέψουμε αυτές τις συνέπειες. Θα ήταν διαφορετικό αν την ένιωθαν την αστάθεια των τιμών οι καταναλωτές, κυρίω με μείωση των τιμών στα καταστήματα. Αλλά στα καταστήματα οι τιμέ δεν αλλάζουν. Όχι μόνο δεν μειώνονται, αλλά αυξάνονται μερικέ φορές. Αλλά δεν νιώθουν αυτή την αστάθεια προς τα κάτω της μείωση των τιμών οι καταναλωτές. Αντίθετα, πλήττονται οι παραγωγοί με αυτή τη μείωση, χωρί κανένα να επωφελείται από αυτό. Και υπάρχουν διαφορές και μεταξύ των κρατών μελών και η διαπραγματευτική ικανότητα μερικές φορές των γεωργών επηρεάζεται από κάτι τέτοιο, γιατί δεν είναι ενωμένοι οι γεωργοί. Και μερικές φορές αποδυναμώνεται η διαπραγματευτική τους ισχύ ακριβώς εξαιτίας της έλλειψης συντονισμού και ενότητας. Ε, αυτή την κατάσταση την εκμεταλλεύεται ο τομέας της διανομής, οι μεγάλες αλυσίδες διανομής. Και εκτός από την αστάθεια των τιμών έχουμε και την κερδοσκοπία. Στην Ευρώπη έχουμε έναν πολύ ασθενή μηχανισμό ρυθμής των τιμών. Και ε, μερικές φορές ε, οι πολυεθνικές έχουν τις ε, έδρες τους σε φορολογικούς παραδείσους και υποφελούνται και ε, από αυτή την κατάσταση. Οπότε είναι σε καλύτερη διαπραγματευτική θέση. Ενώ οι κτηνοτρόφοι και οι γεωργοί μας ε, βρίσκονται σε δινή θέση εξαιτία της αδυναμίας τους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Στην Λετωνία ένα συνέδριο με συμμετοχή άνω των χιλίων γεωργών και κτηνοτρόφων με συζήτηση για το μέλλον και ακόμη και η μεγάλη παραγωγή λαμβάνει το πολύ 15 με 20 σέντ το λίτρο του γάλακτος και είναι ανίκανοι να συμβάλλουν στον προσδιορισμό των τιμών. Και μάλιστα οι τιμές δεν κυμαίνονται πια, έχουν πιάσει πάτο, είναι στο ναδίρ. Δεν επιδέχονται πλέον περαιτέρω διακυμάνσεις. Και ένας από τους λόγους που αντιμετωπίζουν αυτή την καταστροφική κατάσταση οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι μας είναι επειδή σταμάτησαν και εξαγωγές προς τη Ρωσία λόγω του ρωσικού εμπάργου και δεν μπορούν να βρουν εναλλακτικέ αγορές και διεξόδους για τα προϊόντα τους. Αυτή τη στιγμή στην ε, Λιθουανία αντιμετωπίζουμε μεγάλη, μεγάλο πρόβλημα εξαιτία του ρωσικού εμπάργου. Ίσως θα πρέπει να θεσπίσουμε και κάποια συστήματα ασφάλισης του κινδύνου για να δικαιούνται κάποιες ενισχύσεις ε, οι γεωργοί και να ξέρουν ότι είναι εξασφαλισμένο με άλλο το εισόδημά τους. Αλλιώς θα εγκαταλείψουν την Ήπεθρο, θα αφήσουν τα χωράφια τους γιατί δεν βλέπουν πια μέλλον στην Ήπεθρο. Ευχαριστώ κύριος Μποβέ. Ε, ναι, πρώτα απ' όλα ορισμένε παρατηρήσει ε, για τι παρεμβάσει. Κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Όταν είχαμε την μεγάλη αύξηση των τιμών ε, στα ρωσικά σιτηρά, είχαμε ε, μεγάλη κερδοσκοπική δραστηριότητα με πολύ αρνητικό αντίκτυπο. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι ρυθμίζεται από μόνη της αγορά. Υπήρχε σαφής κερδοσκοπική δραστηριότητα από μεγάλο όμιλο συμφερόντων. Και αυτό πρέπει να το επισημαίνουμε γιατί ε, σε τέτοια επίπεδα ισχύω κειμένονται αυτά τα ζητήματα. Μετά, από την 1η Απριλίου και μετά, ε, και τα γαλακτοκομικά προϊόντα εντάσσονται στις χρηματαγορές. Και αυτό μάλιστα από την ημέρα μετά την κατάρριξη των ποσοστώσεων. Επομένω, το να πούμε ότι οι χρηματαγορέ δεν διαδραματίζουν ρόλο δεν ισχύει. Διαδραματίζουν ρόλο και μάλιστα ε, εντείνουν την αστάθεια των τιμών. Είναι ένας παράγοντας που δεν υπήρχε στο παρελθόν, αλλά πλέον ε, είναι εξαιρετικά σημαντικός. Τρίτο και πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το βάρος ε, της διεθνούς αγοράς. Και σήμερα έχουμε όλο και περισσότερο μια λογική συναλλαγματική, όπου το πλεόνασμα των παγκοσμίων αγορών είναι αυτό που προσδιορίζει και την τιμή του γάλακτος. Η τιμή δηλαδή στην οποία βασίζεται και η ευρωπαϊκή τιμή είναι μια αγορά που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα του κόστους παραγωγής. Αυτό ανέφερε το 95 και όπου, ε, με την ευθυγράμμιση των τιμών. Πρέπει λοιπόν να ευθυγραμμίσουμε τους ε, παραγωγούς και την τιμή με ένα κόστος παραγωγής που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και αυτό μας οδηγεί στην καταστροφή, γιατί δεν μπορούμε ε, να ε, το αντιμετωπίσουμε με μία τιμή που να αποσυνδεμένη από Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει ε, να επισημαίνουμε όταν θέλουμε να προτείνουμε λύσεις. Ναι, έχουμε τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής και στο Γάλα είχαμε και είχαμε ψηφίσει στο Κοινοβούλιο. Είχαμε προτείνει λοιπόν να εισαγάγουμε τη δυνατότητα ενίσχυσης των παραγωγών σε περίπτωση υποπαραγωγής και πτώσης των τιμών για να διατηρηθούν τα επίπεδα των τιμών. Και το είχε απορρίψει το Συμβούλιο, να το θυμίσουμε και αυτό, στον τριμερό διάλογο με τη στήριξη της Κομισιόν το είχε απορρίψει. Και έτσι δεν είχε προχωρήσει αυτό το στοιχείο. Σήμερα λοιπόν νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση. Γιατί οι ενισχύσει τη κοινή γεωργική πολιτική δεν βοηθούν καθόλου ε, ω στήριξη του εισοδήματο. Το τμήμα τη κοινή γεωργική πολιτική ε, που ε, στηρίζει τα γεωργικά ε, εργαλεία είναι πολύ μεγαλύτερη, 7-8 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με την ενίσχυση που πραγματικά φτάνει στην τσέπη του γεωργού. Η ενίσχυση λοιπόν έχει ως στόχο την ε, διατήρηση της παραγωγής και δεν αποζημιώνει, δεν σταθεροποιεί τα εισοδήματα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο βλέπουμε ότι ανακύπτει όλο ένα και περισσότερο και στην κρίση την οποία δερχόμαστε σήμερα. Είναι λοιπόν ένα στοιχείο το οποίο θα, μας... θα πρέπει να μας οδηγήσει να πούμε ότι η μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής, γεωργικής πολιτικής δεν ανταποκρίνεται στην κατάσταση των γεωργών και ότι το ζήτημα της σύνδεσης μεταξύ των ενισχύσεων και της στήριξη του εισοδήματο και της παραγωγής είναι κεντρικό ζήτημα. Δεν μπορεί να υπάρξει αποσυνδεδεμένη γεωργική πολιτική. Είναι μία απόλυτη ψευδέστηση ε, που είχε υιοθετηθεί κατόπιν μιας ε, διεθνούς ε, ψευδέστησης και ενός ψευδούς οράματος του ΠΟΕ βλέπουμε και την Αμερική και τον Καναδά που κάνουν διαφορετικά. Μόνο εμείς είμαστε οι καλοί μαθητές που τα εφαρμόζουμε μέχρι το, τα όρια του παραλόγου. Πρέπει λοιπόν να ε, αναθεωρήσουμε αυτή την αποσύνδεση των ενισχύσεων ε, μεταξύ παραγωγής και εισοδών, εισοδημάτων. Αλλιώς δεν θα λειτουργήσει το σύστημα. Σας ευχαριστώ κύριο Σφεράν. Ακούστε. Ασθενίζομαι πλήρως τα σχόλια του προλαλήσαντος. Ε, έχει γίνει έθραυστη και ευάλωτη η Ευρώπη το τελευταίο καιρό. Και ευχαριστώ τους εμπειρογνώμους που προσπαθούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε το ευρωπαϊκό διακύβευμα της γεωργίας, αλλά είναι νοθευμένο το παιχνίδι από την αρχή. Γιατί ε, εδώ και πολύ καιρό βιώνουμε μια περίοδο χαμηλών τιμών και δεν θέλαμε να θυσιάσουμε τη Γεωργία στο βωμό της απελευθέρωσης του, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των Συμφωνιών Ελεύθερων Συναλλαγών. Δυστυχώς σήμερα η Ευρωπαϊκή Γεωργία για μία ακόμη φορά έχει γίνει η μεταβλητή προσαρμογή όλων των πολιτικών προβλημάτων της πολιτικάντικης πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το θύμα αυτής της πολιτικής. Ε, η κατάσταση αυτή οφείλεται σε μία, κατα... σε μία μείωση των τιμών μεταξύ των άλλων προϊόντων και του πετρελαίου που είναι μια βασική πρωτήλη και επηρεάζει την παγκόσμια κατάσταση. Η δραματική κατάσταση που βιώνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Γεωργία δείχνει κάθε μέρα που περνά την επικινδυνότητα της ε, ακρεφνώς ε, φιλελεύθερης πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το μοντέλο αυτό που εδώ και 30 χρόνια μας ε, επέβαλαν οι Βρυξέλλες φάνηκε σήμερα ότι θα πρέπει να το απορρίψουμε. Να αποσυνδεθούμε επιτέλους από αυτό το μοντέλο και να ε, ξεχωρίσουμε τη γεωργία, να στηρίξουμε τους γεωργούς, ώστε κάθε χώρα να ανακτήσει την επισητιστική της κυριαρχία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η εισηγήτρια μας τώρα, η κυρία Ντελαέ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους καλεσμένους ε, εμπειρογνώμονες που ήρθαν να μας διαφωτίσουν ε, η εμπειρία και οι γνώση τους ε, δημιουργούν περισσότερα ερωτηματικά παρά ε, δίνουν απαντήσεις. Και θα ήθελα να με βοηθήσετε όλοι στην εκπόνηση της έκθεσης για να είναι το αποτέλεσμα ενός συλλογικού έργου και όχι η έκθεση μιας μόνο εισηγητήριας. Μιλήσαμε πολύ για τη μεταβλητότητα, την αστάθεια, τι ε, σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών των προϊόντων που οδηγούν στη διακύμανση και του γεωργικού εισοδήματο. Ποια είναι η σχέση τη αστάθειας των τιμών με τη διακύμανση του γεωργικού εισοδήματο. Δεύτερη ερώτηση. Αναφέρθηκε το θέμα των μέτρων διαχείρισης της κρίσης που σήμερα περιλαμβάνονται στον δεύτερο πυλώνα της ανάπτυξης υπαίθρου. Πώς εφαρμόστηκαν αυτά τα μέτρα στα κράτη-μέλη και χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα προγράμματα και όντως συνέβαλαν στη διαχείριση της κρίσης ή στην αναχέτηση της κρίσης. Επίσης κάτι που θα μας βοηθήσει στις ε, μελλοντικές μας εργασίες για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, πώς θα καταπολεμήσουμε μακροπρόθεσμα την αστάθεια των τιμών, αυτή τη μεταβλητότητα στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Κάτι άλλο που επισήμαναν πολλοί εμπειρογνώμονες και το επανέλαβαν και οι συνάδελφοι ε, είναι αν μπορούμε να εμπνευστούμε από τα υφιστάμενα ε, συστήματα ασφάλισης που εφαρμόζουν παγκόσμια εταίροι μας όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες ή ο Καναδάς. Και τέλος, όπως είπε και ο κύριος Ταραμπέλα, συνεχίζονται σήμερα οι διαπραγματεύσεις για το TTIP την διατλαντική εταιρική σχέση. Δεν θα ήθελα να προεξοφλήσω την έκβαση αυτών των διαπραγματεύσεων. Πάντως, στην παρούσα φάση των συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων, πώς ε, θα εντάξουμε το θέμα της καταπολέμησης στάθειας των τιμών στις εμπορικές μας ε, συζητήσεις και σχέσεις ιδιαίτερα στα πλαίσια του TTIP. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ανδριού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ομιλητές για τις παρεμβάσεις τους. Και πάλι δεν υπάρχει κάτι το καινούριο εδώ, γνωρίζουμε την κατάσταση και όλοι εδώ ξέρουμε ότι οι γεωργικές αγορές εκφύσεως δεν είναι σταθερές. Και η κρίση όπως αυτή που περνάμε αυτή τη στιγμή μας το υπενθυμίζουμε. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο λοιπόν ε, να τα σταθεροποιήσουμε. Το φαινόμενο αυτό της αστάθειας έχει ενταθεί τα τελευταία χρονιά και από ε, την νέα κατεύθυνση που έχει πάρει η ευρωπαϊκή αγορά από την απορρίθμιση των αγορών που ξεκίνησε τη δεκαετία του και το υπένθυμισαν ορισμένοι και από την απελευθέρωση των γεωργικών αγορών που ε, συνδέονται και επηρεάζονται από τις διεθνείς συμφωνίες και αυτό υπόθηκε. Αυτή η αστάθεια των τιμών είναι ένα επικίνδυνο φαινόμενο από πολλέ πτυχές. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την επιστημιστική ασφάλεια. σε ό,τι φορά δηλαδή την δυνατότητα του καταναλωτή να ε, τραφεί. Μετά και για τους παραγωγούς είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί πρέπει να δοθεί και μία προοπτική στους γεωργούς ε, επιβίωσης ε, και εξυγχρονισμού τους. Και μετά και για τις επιχειρήσεις ε, του επιστημισμού γιατί πρέπει και αυτές να έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. Είναι απαραίτητο λοιπόν να επενθυμίσουμε την ε, καλύτερη ρύθμιση στις γεωργικές αγορές. Δεν μπορούμε να ξεχνούμε ότι οι μεγάλες περιφέρειες του κόσμου, το αναφέραμε και αυτό στο προηγουμένως, ότι έχουν ε, γεωργικές πολιτικές για τη διασφάλιση της επιστημιστικής ασφάλειας και ε, για να μην εξαρτώνται πλήρως από το εξωτερικό για την ε, κάλυψη των γεωγραφικών του αναγκών. Αναφέρθηκε αυτό και για την ΕΠΑ και για αλλού. Πρέπει να το θέτουμε παράλληλα και με προπολογισμού και άλλα στοιχεία. Ο προπολογισμό τη ΕΚΑΠ είναι 38% ε, του προπολογισμού, ενώ είναι μόλις 1% των προπολογισμών που, των κρατών μελών. Επομένως βλέπουμε και την πολιτική βούληση που υπάρχει για να έχουμε μια πραγματική ε, πολιτική δυναμική. Και νομίζω ότι αυτή η ρύθμιση θα πρέπει να τεθεί στο πλαίσιο της κοινή γεωργικής πολιτικής με δημόσια ρύθμιση για παρέμβαση αρχικά Ο Επίτροπος ε, νομίζω ότι κάτι θα έχει αποκομίσει από την κατάσταση που ε, εξετάζουμε σήμερα. Δεν πρέπει να επανέλθουμε στις παρεμβάσεις του παρελθόντος, όμως να εφαρμόσουμε νέα, πιο προσαρμοσμένα μέτρα ε, στη σημερινή κατάσταση, αλλά και ιδιωτική παρέμβαση στήριξη στην διάρθρωση των ε, κλάδων. Όμως θα πρέπει να συμπληρωθεί αυτή η ρύθμιση και με διεθνείς κανόνες και πρότυπα που θα έχουν ως στόχο να περιορίσουν την ε, κερδοσκοπία στις ε, πρώτες ύλε και τα ε, τρόφιμα για να ενισχύσουμε τη σταθερότητα των αγορών. Και τώρα θα ήθελα να θέσω τα εξή ερωτήματα στους ομιλητές μας. Μπορούμε να πούμε ότι η αστάθεια των τιμών στις πρώτες γεωργικές ύλε έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. συχνά τίθεται αυτό το ζήτημα. Μπορούμε να εκτιμήσουμε την έκταση του φαινομένου της κερδοσκοπίας στις ε, γεωργικές αγορές και τέλος τι είδους ρύθμιση θα μπορούσαμε να έχουμε. Άκουσα τα όσα είπαν ε, και από το Πανεπιστήμιο της Γάνδης. Δηλαδή να βρούμε ε, μια τροχοπέδη για, την, για τον περιορισμό της παραγωγής. Έχει ενδιαφέρον αυτή η πρόταση, αλλά τι είδου ρύθμιση θα μπορούσαμε να εισαγάγουμε σήμερα στην κοινή γεωργική πολιτική όπως έχει σήμερα, αλλά και στη μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2020. Ευχαριστώ κύριε Ζιάρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πάρα πολύ και, πάρα πολύ και τους εμπειρογνώμονες ε, συμφωνούμε όλοι μας ότι δεν πρόκειται για ε, κανονικές διακυμάνσεις τιμών, αλλά πρόκειται για το ότι οι τιμές έχουν φτάσει σε ένα κατώτατο όριο ε, που διαρκεί καιρό και ένα όριο το οποίο απλά θέτει σε κίνδυνο την χρηστή διαχείριση και αποτελεσματική διαχείριση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Υπάρχουν πολλά πράγματα που με καθιστούν δίβουλο. Εγώ μεγάλωσα, ξέρετε, σε ένα σύστημα όπου υπήρξαν, υπήρχαν ρυθμίσεις για τις ποσότητες, υπήρχε κεντρικά κατευθυνόμενη οικονομία, το πόσο μπορούσαν και έπρεπε να παραχθεί, υπήρχαν και εγγυμένες τιμές, αλλά παρόλα αυτά το σύστημα απέτυχε. Και θέλω να κάνω τρεις ερωτήσεις. Θεωρώ το θέμα σωστό. Η πρώτη μου ερώτηση λοιπόν είναι η εξή. Έχετε μήπως μία ιδέα για το ποια θα πρέπει να είναι η σχέση ανάμεσα στην ενίσχυση με βάση το δικό σας μοντέλο και την ίδια ευθύνη των επιχειρηματικών των επιχειρηματιών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Δεύτερη ερώτηση. Έχετε μια ιδέα ε, το ποιοι είναι οι πόροι που χρειαζόμαστε για το ένα ή το άλλο μοντέλο. Ε, είναι αλήθεια ότι κάποια στιγμή ε, χρειαζόμαστε χρήματα για να χρηματοδοτήσουμε αυτό το σύστημα. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι ένα ερώτημα το οποίο αφορά μόνο τη Γερμανία έχουμε το εξής πρόβλημα. Η ε, αυτάρκεια στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ε, είναι πολύ δύσκολη. Η αστάθεια των τιμών σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν και κάποιες καλές χρονιές, αλλά τελικά είναι πάρα πολύ δύσκολο οι γεωργοί ε, σε καλές χρονιές να μπορέσουν να δημιουργήσουν κάποιο οικονομικό απόθεμα. Και γι' αυτό οι γεωργοί δεν έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν κάποιες ευθύνες. Μήπως θα πρέπει και αυτό να το λάβετε υπόψη σας στα μοντέλα που μας παρουσιάσατε. Ευχαριστώ κύριε Στεκάστρο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συγχαρητήρια στην ομάδα των εμπειρογνωμόνων γιατί μας παρουσίασαν θέματα πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα για τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Νομίζω ότι έχει έρθει η στιγμή όπου το Κοινοβούλιο, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, ε, θα έπρεπε να κάνει κάποιες αλλαγές, αλλά δεν τις έκανε. Η αστάθεια των τιμών είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, ε, το οποίο δημιουργεί δυσκολίες στις επιχειρήσεις, κυρίως ε, στη διαχείριση των επενδύσεων και θέλω να ρωτήσω κάτι ξεκάθαρα τους εμπειρογνώμονες. Κοιτάξτε, εν ώψη της ακαμψίας ε, του οικονομικού προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς μπορούμε να εισάγουμε εργαλεία όπως είναι οι αντικυκλικές ε, πληρωμές ή μηχανισμοί διαχείρισης της αστάθειας των τιμών, παρότι όπως σας λέω υπάρχει μια χρηματοψηφιακή ακαμψία. Ας το πω αλλιώς, πώς μπορούμε συγκεκριμένα να προτείνουμε τι μπορούμε συγκεκριμένα να προτείνουμε χωρίς να αλλάξουμε τα χρηματοψηφιακά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί αυτό έχει μια πολύ μεγαλύτερη δυναμική από αυτήν με την οποία μπορούμε εμείς σήμερα να ασχοληθούμε. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πάρα πολύ τους εμπειρογνώμονες για τις παρεμβάσεις τους. Και εγώ είμαι λιγάκι δίβουλος, αμφιταλαντεύομαι για το ποιο είναι το σωστό σύστημα. Είχαμε ανώτατες τιμές στο γάλα και παρόλα αυτά 30 μέχρι 40 σεντ ε, διακυμένονται οι τιμές ε, για το προϊόν αυτό. Τώρα, εφόσον μιλάμε για το ότι θα πρέπει πάλι να επανεισάγουμε το σύστημα του ελέγχου ποσοστώσεων, θα ήθελα να μας πούνε οι εισηγητές ποιο σύστημα τελικά είναι αποτελεσματικό. Μπορείτε να φανταστείτε στην Ευρώπη να υπάρχει ας πούμε στο γάλα ένα πανευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου παραγωγής και αν ναι θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα στο σύνολο της Ευρώπης. Το τρίτο, ε, τιμή παρέμβασης. Σήμερα υπάρχει στην αγορά και νομίζω ότι το σύστημα αυτό στο γάλα περισσότερο βλάπτει παρά ωφελεί το γάλα. Ε, γιατί σας λέω ότι η τιμή του γάλακτος είναι πάνω από την τιμή παρέμβασης. Αυτή τη στιγμή το γαλακτοκομείο μπορεί να έχει 29 σεντ και η τιμή παρέμβαση είναι 22, άρα δεν συμφέρει. Γι' αυτό λοιπόν Βεβαίως και τα πράγματα ποικίλουν στα κράτη-μέλη, αλλά εμείς θα θέλαμε να ασκήσουμε πίεση. Ε, εγώ ήθελα να ε, συντάξω την έκθεσή μου και να πω ότι πρέπει να ασκήσουμε πίεση τα κράτη-μέλη όσον αφορά το φορολογικό. Ε, περάσανε πολλά χρόνια όπου οι γεωργοί είχαν καλά αποτελέσματα, αλλά τότε ξέρετε το 45% του κέρδους τους το απέδωδαν στο κράτος. Επειδή όμως η γεωργία εξαρτάται άμεσα από το κλίμα και από άλλους παράγοντες, πρέπει οι γεωργοί να έχουν απόθεμα οικονομικό για κακές χρονιές για χρόνια κρίσης. Αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να το θίξουν οι κύριοι καθηγητές. Και το τελευταίο, θέλω να πω πραγματικά συγκλονίστηκα για το πόσο πολύ εκμεταλλεύεται το εμπόριο, την ε, εξουσία του στην αγορά. Μία, ένα γαλακτοκομείο μου είπε ότι η τιμή των τηλεκομικών προϊόντων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τιμή του γάλακτος. Στην Γερμανία υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση του εμπορίου και με εξέπληξε που ένας σοσιαλδημοκράτης υπουργό Οικονομικών σε αντίθεση με το ομοσπονδιακό, ε, την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Καρτέλ, σε αντίθεση με την Βέρντι τελικά επέτρεψε να λειτουργήσουν δύο τόσα μεγάλα ολιγοπόλια στη Γερμανία. Ε, το να το κάνει αυτό ένας φιλελεύθερος θα το καταλάβαινα, αλλά ένας σοσιαλδημοκράτης πραγματικά με εξέπληξε. Μάλιστα. Δεν ε, ζητά άλλος κανείς το λόγο σε αυτό το γύρο. Αν μου επιτρέπετε, θέλω και εγώ να υποβάλω μια ερώτηση οι δοκιμάσεις των τιμών συνδέονται και με τις ιδιαιτερότητες της γεωργίας που επηρεάζεται από τις μετεωρολογικές συνθήκες, από τις καιρικέ συνθήκες που επηρεάζουν και τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Αυτές οι διαφορές βρίσκονται στο DNA της γεωργίας. Επίσης, ε, έχουμε τρεις διαδοχικές πενταετίες ε, με διαφορετικές σχέσεις και είναι κάπως φυσιολογικό. Ε, στις διαδοχικές τριετίες ε, άλλοι τομείς ενισχύονται και άλλοι αποδυναμώνονται. Έχουν άνθηση και παρακμή. Επίσης, σε παγκόσμια κλίμακα ακριβώς επειδή έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση στις ε, παγκόσμιες αγορές και λόγω του ανοίγματο ε, και της παγκοσμιοποίησης θα περιμέναμε θετικά αποτελέσματα. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και αρνητικά και το άνοιγμα των παγκόσμιων αγορών ε, επηρεάζει αρνητικά τα επίπεδα των τιμών. Διακοιμάνσεις έχουμε και στην παραγωγή. Βέβαια, για την παραγωγή δεν είναι αρμόδιος μόνο ο Γιώργος. επηρεάζεται και από πολλούς εξωτερικούς παράγοντες στο επίπεδο της παραγωγής του. Όλα αυτά συμβάλλουν ε, στο φαινόμενο της αστάθειας. Λοιπόν, τώρα ο λόγος και πάλι στους εμπειρογνώμονες. Ε, δεν χρειάζεται να λάβετε όλο το λόγο αν θεωρείτε ότι δεν αφορούσαν εσάς τα σχόλια ή οι ερωτήσεις. Δύο λεπτά ο καθένας και τρεις παρακαλώ εμπειρογνώμονες σας λάβουν το λόγο, όχι περισσότεροι. Παρακαλώ. Με τη σειρά που μιλήσατε και προηγουμένως, ο κύριος Φερέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από τις παρεμβάσεις που ακούσαμε διαπιστώνουμε ότι το πρώτο πρόβλημα της αστάθειας είναι πολιτικού χαρακτήρα. Αν σήμερα έχουμε αστάθεια και μεταβλητότητα στις τιμές, αυτό οφείλεται στο άνοιγμα των αγορών, που είναι απόρρια των ε, ηλιμένων ε, δεσμεύσεων. Και η εφαρμογή τεχνικών λύσεων στην κατάσταση αφορά και, την, ε, και το διεθνές πολιτικό κλίμα και περιβάλλον και το κατά πόσο θα το αλλάξουμε, γιατί έχουμε υπογράψει συγκεκριμένες συμφωνίες, έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. Και μερικές από αυτές τις δεσμεύσεις και τις συμφωνίες μας απαγορεύουν να χρησιμοποιήσουμε ε, συγκεκριμένα μέσα και μηχανισμούς. Οι διακυμάνσεις τιμών δεν σημαίνει και αστάθεια τιμών. Οι διακυμάνσεις είναι φυσιολογικές. Η αστάθεια είναι ε, μεγάλη μεταβλητότητα, μεγάλες μεταπτώσεις και ο χαρακτήρας της αβεβαιότητας ταυτόχρονα. Αλλά η διαδικασία είναι αμφίδρομη. Γιατί μερικές φορές συνδέουμε το, τη λήξη των ποσοστώσεων με την έναρξη της αστάθειας. Αυτό δεν ισχύει. Το 2008-2009 είχαμε στο γαλακτοκομικό τομέα ε, με απότομες αυξήσεις τιμών και απότομες μειώσεις. Ενώ είχαμε ποσοστώσεις. Γιατί, γιατί η κοινή γεωργική πολιτική δεν είναι πια ένα πάνεμο λιμάνι. Βρισκόμαστε στα μέσα του ωκεανού και μάλιστα αντιμετωπίζουμε και καταιγίδε. Οι διεθνείς τιμές έχουν φτάσει τώρα και στις ευρωπαϊκές αγορές. Και από αυτές επηρεαζόμαστε. Βέβαια, δεν επηρεάζονται όλα τα προϊόντα με τον ίδιο τρόπο. Μιλούμε για τα βασικά προϊόντα, μιλούμε ε, για τα σιτηρά, τα γαλακτοκομικά, τη ζάχαρη, αλλά δεν καλύπτονται από το φαινόμενο αυτό όλα τα γεωργικά προϊόντα. Δεύτερον, αν εφαρμόσουμε τα ίδια κριτήρια, είναι σαφές ότι για τα μεγάλα προϊόντα έχουμε υποστεί την αστάθεια των τιμών. Ας μην ξεχνούμε ότι οι τιμές των σιτηρών καθορίζονται στη Βόρεια Αμερική για τον κόσμο. Ενώ τα... οι τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων καθορίζονται στην Αυστραλία. Αν μειώσουμε τον όγκο παραγωγής με δραστικό τρόπο για να αυξηθούν οι τιμές, οι, οι παγκόσμιες τιμές θα αυξηθούν, όχι οι ευρωπαϊκές τιμές μόνο. Οπότε ποιοι θα έχουν κερδισμένοι, οι υπόλοιποι, όχι εμείς. Και αν εμείνουμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που σέβεται τις συμβάσεις που έχει υπογράψει, τις συνθήκες που έχει ε, συνομολογήσει και τους κανόνες που έχει ασθενιστεί, νομίζω ότι είναι απαραίτητο όχι να θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την αστάθεια και να παίζουμε με αυτή, αλλά να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τους παραγωγούς από την αστάθεια αυτή. Δεν είναι το ίδιο. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους γεωργούς, τους παραγωγούς μας. Και αν θέλουμε να τους προστατεύσουμε, εγώ βέβαια ένα σύστημα μόνο γνωρίζω που ε, απαλλάσσει από τους κινδύνους και το σύστημα αυτό είναι το ασφαλιστικό, οι ασφαλίσεις. Και η κοινή γεωρική πολιτική της περίοδου 2014-2020 επιτρέπει στο δεύτερο πυλώνα τη θέσπιση ασφαλιστικών συστημάτων που μπορούν να εφαρμοστούν, επιτρέπονται μάλιστα και οι μεταφορές μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα στα πλαίσια των κονδύλιων που έχουν τα κράτη-μέλη και των σχετικών προϋπολογισμών. Επίσης, ε, ε, τι καθορίζει ε, τη βιωσιμότητα ενός παραγωγού, το περιθώριό του και όχι το εισόδημά του. Ας αφήσουμε τη συζήτηση για το εισόδημα και περιοριστούμε στη συζήτηση για το περιθώριο. Αυτή καθορίζει τη βιωσιμότητα μιας γεωργικής εκμετάλλευσης. Ευχαριστώ. Ehm, και εγώ θα είμαι πολύ σύντομος. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Νομίζω είναι σαφές ότι παρουσιάσαμε πως η αστάθεια των τιμών είναι ένα πολύ περίπλοκο φαινόμενο. Υπάρχουν ε, διάφορες μακροοικονομικές ε, μεταβλητές, ε, ισοτιμίες, η σχέση με άλλες τιμές. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε την αστάθεια και πώς θα μπορεί κανείς να διαχειριστεί μία γεωργική αγροτική εκμετάλλευση έτσι ώστε να ε, περιοριστούν ε, τα στοιχεία της αστάθειας. Νομίζω λοιπόν ότι το θέμα του περιορισμού της ε, παραγωγής, παρότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, πρέπει να εμβαθύνουμε σε αυτό. Από τη μια έχει τους περιορισμούς ε, που είπε ο συνάδελφος, δηλαδή είμαστε σε ένα παγκόσμιο, σε μια παγκόσμια αγορά και δεν έχουμε μόνο την ευρωπαϊκή να αντιμετωπίσουμε. Από την άλλη υπάρχει η ακαμψία της ε, προσφοράς. Ε, αυτό είναι σαφές, διότι η γεωργία είναι ένας παραγωγικός κύκλος ε, που ξεκινάει σε μια συγκεκριμένη περίοδο και τελειώνει επίσης σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Κατά τα άλλα έχουμε κάνει κάποιους πειραματισμούς με το γάλα, το θέμα του, των τραστ ε, δεν είναι εύκολο να το διαχειριστεί κανείς ε, κυρίως για ορισμένα προϊόντα γιατί υπάρχουν αρκετές ιδιαιτερότητες. Όσον αφορά το θέμα του καταναλωτή, ε, εντάξει δεν είχαμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας αλλά νομίζω επισημάναμε πως ο μηχανισμός της αστάθειας των τιμών δεν είναι επαρκής. Είδαμε πως το θέμα της διαφάνειας είναι καθοριστική σημασία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Διαφάνεια λοιπόν θέμα πολύ μεγάλη σημασία και κλείνω με μία παρατήρηση. Τα ε, εργαλεία τα οποία είναι σημαντικά για να λειτουργήσει η Ευρώπη, ε, για να δούμε πώς ο Γεωργός μπορεί να διαχειριστεί την αστάθεια των τιμών στο εισόδημά του, νομίζω ότι αυτό ήταν μία σωστή τοποθέτηση του θέματος. Υπάρχει το θέμα των αποθεμάτων, αυτό που είπε και ο κύριος Δες, οικονομικά αποθέματα αποταμιεύσεις δηλαδή, το να δώσει κανείς ε, τη δυνατότητα στον ε, Γιώργο να έχει αποταμιεύσεις χωρίς αυτές να υπόκεινται σε φορολογία, αυτό σημαίνει θα μπορούσε να υπάρχει ένας ειδικό λογαριασμός και εκεί να βάζει ο Γεωργός τις αποταμιεύσεις του έτσι ώστε να τις χρησιμοποιήσει όχι μόνο όταν θα υπάρχουν οι κρίσεις της αγοράς ε, που θα φέρνει το εισόδημα κατά 70% πιο κάτω, αλλά και για να μπορέσει μακροπρόθεσμα να αντιμετωπίσει μικρές ζημιές. Γιατί ο Γιώργος αντιμετωπίζει τέτοιες μικρές ζημιές. Είναι μακρύς ο κύκλος της ε, παραγωγής, ε, χρειάζεται κεφάλαιο, άρα λοιπόν να υπάρξουν διάφορα προγράμματα. Σε κράτη-μέλη έχουν υπάρξει πρωτοβουλίες. Η εμπειρία του Καναδά μας δείχνει το εξής. Καλύτερα παρεμβάσεις αντικυκλικές, ε, ακόμα και αν υπάρχει ο κίνδυνος έλλειψης διαφάνειας, γιατί αυτό σημαίνει ότι ε, υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό και ο ε, γεωργός όταν θέλει να κάνει μια επένδυση μπορεί να καταφύγει σε αυτό το κεφάλαιο το ε, εργαλείο αυτό της αποσταθεροποίησης είναι κάτι το οποίο μοιάζει λιγάκι, αλλά ε, το θέμα είναι ότι σε αυτό το εργαλείο που αναφέρεται έχουμε μία εκ των υστέρων ε, παρέμβαση, ενώ στην παραδοχή που εκφράζουμε εμείς ή εκφράζω εγώ είναι η παρέμβαση γίνεται εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων. Σήμερα ρώτησε κάποιος ε, ποια είναι τα χρήματα, οι πόροι που επενδύει επενδύει η Ευρώπη. 3,3 δις για αυτά τα εργαλεία σταθεροποίησης. Αυτό είναι το ποσό. Περίπου 3,3 δις. So there a couple of Υπήρξαν ορισμένα ερωτήματα σε ό,τι αφορά τον περιορισμό της ε, ποσότητας και να ξεκαθαρίσω ότι δεν θεωρώ ότι πρέπει να επιστρέψουμε στην περίοδο των ποσοστώσεων γιατί όπως ανέφεραν πολλοί ευρωβουλευτές και την περίοδο των ε, ποσοστώσεων υπήρχε αστάθεια ε, στις τιμές. Απλώς κάνω την αντιστοίχηση με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στο παρελθόν είχαμε κάτι αντίστοιχο με ορισμένε χώρες. Ε, η υποχρέωση του ΣΕΤΑΣΑ της αποθήκευσης της αγανάπαυσης, συγγνώμη, υπήρχε στο παρελθόν, αλλά αυτό δεν εφαρμοζόταν τυχαία, εφαρμοζόταν σε περιόδους ε, υψηλών τιμών. Στην στο Αμερικανικό πρόγραμμα σε ό,τι αφορά την, ε, την διατήρηση του ορίου υπήρχε αρχικά σε πραγματεύσεις, αλλά όχι τελικά. Όταν λαμβάνουν οι γεωργοί ενισχύσεις θα περιόριζαν και την ε, παραγωγή τους. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένα τέτοια παραδείγματα. Και συμφωνώ ότι αυτό δεν θα έχει τεράστια επίπτωση ε, στην τιμή, γιατί είναι μεγάλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν έχει μεγάλο αντίκτυπο στην παγκόσμια αγορά στην οποία συμμετέχει και δεν μπορούμε να πω ακριβώς ότι αυτή είναι η χρυσή τομή. Αναφέρω απλώς ότι μπορούμε να το, μπορείτε να το εξετάσετε και μπορούμε να αναζητήσουμε παραδείγματα που ε, λειτουργήσαν θετικά στο παρελθόν ε, και στην γεωργική πολιτική αλλά και στην, στον τομέα της ηλεκτρικής ε, ενέργειας. Τώρα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του τρέχοντος πυλώνα 2 και των μέσων που διατίθεται εκεί, πολύ λίγα κρατημέλη ε, πήραν την πρωτοβουλία να το υλοποιήσουν. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν είναι εύκολο να ενθαρρύνουμε τον ιδιωτικό τομέα, ακόμα και με τη δημόσια στήριξη, να συστήσουν τέτοια προγράμματα ασφάλισης. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό που έχουν εξεταστεί ενδελεχώς επιμέρους ε, μελέτες. Κάποιος ανέφερε το ζήτημα της ισχύω της αγοράς και της ε, πτυτικότητας, της αστάθειας, Όντω θα μπορούσαν να υπάρχουν ζητήματα του market power, όμω εκεί υπήρξε και αναφορά και στον τομέα των γαλακτοκομικών. Εγώ νομίζω ότι αυτό ο κλάδο είναι εκεί όπου οι συνεταιρισμοί έχουν μεγάλο μερίδιο τη αγορά. Αλλά ακόμα και αυτό, από ό,τι φαίνεται, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και να λύσει το θέμα τη αστάθεια. Επομένω, το να εξετάσουμε μόνο την ε, ισχύ τη αγορά ω μοναδική λύση για να επιλύσουμε την αστάθεια δεν ισχύει. Και τέλος, για να μην υπερβώ και το χρόνο μου παραπάνω, για την τελευταία παρέμβαση, όντως θεωρώ ότι η αστάθεια ενέχεται στην γεωργική παραγωγή. Το γνωρίζουν και, και οι ίδιοι οι παραγωγοί, οι αγρότες. Το θέμα είναι σε, σε ποιο βαθμό μπορούν να βοηθήσουν και οι υπεύθυνοι χάραξη πολιτικής. Uh, so many uh, πολλές ε, ερωτήσεις υπευλήθησαν. Δύσκολο είναι να τις καλύψουμε σε μία μόνο απάντηση θα επικεντρωθώ σε ορισμένα θέματα. Η αστάθεια είναι ο τρόπος αγοράς να σας πει αν θέλει ένα προϊόν ή όχι. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε έναν τρόπο στον κόσμο να ελέγχει τις τιμές. Επίσης, δεν μπορούμε να ελέγξουμε την αστάθεια των τιμών με τις ποσοστώσεις. Είδαμε ότι αυτό δεν λειτουργεί. Γιατί για το αποπτυρωμένο γάλα σε σχόλιο υπάρχει ένα σύστημα ποσοστώσεων, αλλά τελικά ποιο είναι το αποτέλεσμα. Οι Αμερικανοί παραγωγή πουλάν σε χαμηλότερες τιμές από τους Ευρωπαίους. Ουσιαστικά δηλαδή με το σύστημά μας βοηθούμε τους Αμερικανούς να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην ευρωπαϊκή αγορά. Θα πρέπει επίσης να διαχειριστούμε τη, το, το κίνδυνο και την αστάθεια των τιμών. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε βρει κατάλληλους μηχανισμούς θα πρέπει να έχουμε μηχανισμούς να ελέγξουμε τις, ε, τις ποσότητες των προϊόντων και κάποιες, κάποια, κάποιες δείκτες τιμών ίσως θα πρέπει να ληφθούν ώστε όταν ε, είναι 40 λεπτά, 40 λεπτά το λίτρο και φαίνεται να μειώνεται να μην ε, επενδύουν σε αύξηση της παραγωγής θα πρέπει να λαμβάνουμε ως ε, σημάδια τις, τις τάσεις των δημών. Επίσης, ε, για πρώτη φορά ε, μέσα 25 χρόνια μας λένε πόσο μπορούμε να παράγουμε και ποιος θα είναι ο ποιος, ποιες θα είναι οι τιμές του γάλακτος. Τεράστιες οι διαφορές σε σχέση με πριν από 25 χρόνια. Κατάλαβα αυτά που είπε ο κύριος Ροπέ σε ό,τι αφορά την απερίμωση της υπαίθρου. Όντως δεν υπάρχουν κίνητρα, αλλά εγώ δεν θα μπορούσα να είχα παραμείνει στην φάρο μου και η αδερφή μου το ίδιο, αν η πολιτική δεν είχε αλλάξει και αν έμενε στα παλιά. Γιατί είχαμε πολύ μικρή γεωρική εκμετάλλευση. Τώρα έχουμε μεγαλύτερη ευκαιρία από ποτέ να αυξήσουμε την παραγωγή, να αυξήσουμε τα κοπάδια μας και να βελτιώσουμε τις επιχειρήσεις μας. Τώρα έχουμε καλύτερες ευκαιρίες ε, γιατί η επιχείρηση είναι σε τελική ανάλυση που θα πρέπει να, λάβε, να λαμβάνετε υπόψη και δεν είναι μόνο πολιτικό το θέμα. Οπότε θα πρέπει πάνω απ' όλα να εξασφαλίσουμε την δυνατότητα των γεωργών να παραμείνουν στις εκμεταλλεύσεις τους. Όντως, πολλές ερωτήσεις ε, ε, διατυπώθηκαν και αυτό δείχνει το ζωηρό ενδιαφέρον για το πρόβλημα που είναι όντως πολύ σπουδαίο. Όπως είπε ο κύριος Μποβέ, η σημερινή κυνηγιορική πολιτική σχεδιάστηκε στα πλαίσια των εξελίξεων στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου, που δεν εξυπηρετούσε κατά ανάγκη την επισητιστική ασφάλεια, αλλά στήριζε περισσότερο τη γεωρική παραγωγή. Υπήρχαν άλλα κίνητρα που τότε ήταν εύλογα, αλλά σήμερα δεν μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε τις διαδοχικές κρίσεις. Και πέραν της αστάθειας των τιμών έχουμε και το άνοιγμα των παγκόσμιων αγορών. Και όπως είπαν ε, κύριε Δεκάστρο και κύριε Ζιά, πώς είναι δυνατόν με τον προπολογισμό μας να αντιμετωπίσουμε αυτό το μείζον πρόβλημα της αστάθειας των τιμών. Πάντως ε, πιστεύω ακράδαντα ότι παρόλα αυτά μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, αλλά θα πρέπει να κάνουμε καλύτερο επιμερισμό των διαφόρων πτυχών της γεωργικής πολιτικής. 60% του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Προϋπολογισμού αφιερώνεται σε αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις. Βέβαια αυτό εξηγείται από τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου και μάλιστα όταν οι ψηλές οι τιμές είναι αποσυνδεδεμένες δεν, δεν, δεν βοηθάν και το ίδιο όταν είναι και χαμηλές οι τιμές. Υπάρχουν κίνδυνοι που ξεπερνούν κατά πολύ ε, τους κινδύνους που μπορεί να διαχειριστεί ο κάθε γεωργό. Αυτό θα πρέπει να επανέλθουμε σε μια ε, γεωργική πολιτική που πάνω απ' όλα θα εφαρμόζει και αντικυκλικές ενισχύσεις οι οποίε θα είναι καλά πλαισιωμένε. Γιατί αν θέλουμε να διαχειριστούμε αυτό το άνοιγμα προ τι παγκόσμιε αγορέ, θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον κάποιε δράσει για να αντιμετωπίσουμε είτε τι πολύ υψηλέ είτε τι πολύ χαμηλέ τιμέ. Και θα πρέπει να κάνουμε και μία ιεράρχηση των δράσεών μας. Είτε των δράσεων που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό, είτε από τον εθνικό υπολογισμό, είτε από τους κλαδικούς προϋπολογισμούς. Και θα πρέπει να κάνουμε μια σωστή ιεράρχηση. Επίσης μιλήσαμε για τα ασφαλιστικά συστήματα. Φυσικά δεν είναι παντοδύναμα αυτά τα ασφαλιστικά συστήματα και δεν μπορούν να λύσουν όλα τα προβλήματα. Θα πρέπει φυσικά να έχουν κάποιε εξασφαλίσει για το περιθώριό του οι γεωργοί, αλλά δεν πρόκειται να ασφαλίσουμε το ε, περιθώριο αν δεν καταπολεμήσουμε στι στις ανοιχτές αυτές παγκοσμιωμένες αγορές ε, το φαινόμενο της αστάθειας των δημών. Δυστυχώ δεν μπορώ να επεκταθώ περαιτέρω γιατί εξάντλησα το δίλεπτο. Μίλησα για δυόμιση λεπτά για την ακρίβεια. Μάλιστα. Στο πρώτο σκέλος ασχοληθήκαμε με την παρούσα κατάσταση, τώρα θα περάσουμε στις μελλοντικές προοπτικές. Θα ήθελα στο δεύτερο γύρο να επικεντρωθείτε κυρίως ε, σε υποβολή ερωτημάτων προς τους ε, εμπειρογνωμονές μας. Μελλοντικές προοπτικές λοιπόν. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον κύριο Φέντον για 8 λεπτά. Thank you. Ευχαριστώ. This is the usual. I represent a financial. Εκπροσωπώ ε, μια εταιρεία οικονομικών ε, υπηρεσιών. Βρισκόμαστε στην, στο κατάλογο Fortune 500 ε, και είμαστε μία οντότητα που ρυθμίζεται πλήρως από τις αρμόδιες αρχές, ε, το, τις Αμερικανικές και το ε, τα αναφέρω αυτά πάντοτε, κάνουμε μια παρουσίαση εξ ονόματος της ε, επιχείρησης. Μία σύντομη ε, εισαγωγή για το ποιοι είμαστε, την αστάθεια των τιμών των γαλακτομικών, τα είπαμε βεβαίως αυτά, ε, Πώ ακριβώ διαχειριζόμαστε αυτή την αστάθεια στην Αμερική, αν αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει στην Ευρώπη ε, και πώς μπορούμε να αναπτύξουμε στην Ευρώπη ε, συμπεράσματα. Είναι τεχνικό το ζήτημα, δεν έχω και πολύ χρόνο. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να διευκρινίσω ορισμένα ζητήματα στα οποία θα ήθελα να σταθώ για ένα συγκεκριμένο κλάδο. Η INTL FC Stone Dairy ασχολείται με τη διαχείριση κινδύνων στα γαλακτομικά. Ασχολούμαστε με εργαλεία που αξιοποιούνται ε, στο 90% και στην Ευρώπη. Και ε, συμμετέχουμε και στην αγορά, την προθεσμική αγορά στη Νέα Ζηλανδία, ε, αλλά και στην Αμερική. Επόμενη διαφάνεια. Εδώ έχετε μια εικόνα της γεωγραφικής μας δραστηριότητα. Και αυτό ήθελα να αναφέρω ότι είναι θέμα περιθωρίου και όχι διαχείρισης ε, τιμών. Την ίδια αρχή έχουμε και σε ό,τι αφορά τη δοσοκομεία, τα γαλακτομικά, όλα τα προϊόντα. Τώρα, πόσο, πόση αστάθεια υπάρχει στα γαλακτοκομικά για να σας το εξηγήσω με μεγαλύτερη, σε μεγαλύτερο βάθος. Εδώ βλέπετε αυτή τη διαφάνεια, στο κάτω μέρος έχουμε το, το χρόνο, Γενάρης του 2002, Γενάρης του 2017 και στον κάθετο άξονα έχουμε την μεταβολή των τιμών σε ποσοστό. Βλέπετε λοιπόν ότι είμαστε συν 10 πλην 10% κατά κύριο λόγο. Ε, μιλούμε για μία περίοδο 4 και 12 εβδομάδων. Η κόκκινη γραμμή είναι αυτή με τις 4 εβδομάδες. Βλέπετε λοιπόν ένα πραγματικό γράφημα της S&P που είναι ε, το χρηματιστήριο. Όλοι ξέρουμε πώς η αστάθεια υπάρχει και, και ε, ευμεταβλητότητα υπάρχει στο χρηματιστήριο και πόσο μπορεί κάποιος να χάσει, να κερδίσει ανάλογα με τις μεταβολές στο χρηματιστήριο. Βλέπετε λοιπόν ότι αυξήθηκε η μεταβολή ε, κατά τη διάρκεια της πιστοτικής κρίσης ε, από το 2008 μέχρι το 2010. Η αστάθεια από το σύνηθε 10% πάνω κάτω, ε, συμπλήν δηλαδή, πήγαμε στο 20 συμπλήν. Και θυμάστε και στον τύπο που ακούγαμε την υψηλότερη αστάθεια για πόσο τρομερή εποχή ήταν εκείνη. Τώρα επόμενη διαφάνεια. Βλέπετε εδώ το αντίστοιχο γράφημα για το αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη από τον Γενάρη του 1990 μέχρι τον Γενάρη του 2000. Και εδώ βλέπετε ότι η μεταβολή των τιμών είναι πάλι στην πλήν 10%. Είναι ένα αρκετά ήπιο, ας πούμε, προϊόν με ήπια μεταβολή. Εδώ έχετε ένα γράφημα της, του αποβουτυρωμένου γάλακτος σε σκόνη και πάλι από το 2000 μέχρι το 2017. Και εδώ βλέπετε ότι ήταν σαν να, σαν να έπαθε καρδιακό επεισόδιο ο ασθενής εντό εισαγωγικών. Από το σύν 10% πήγαμε μέχρι και συν 40 πλήν 30%. Καμία σχέση δηλαδή με αυτό που σας έδειξα προηγουμένως. Τελικά λοιπόν ποιος ε, προσπάθησε να αντιμετωπίσει αυτή την αστάθεια, αφενός ο παραγωγός από τη μία πλευρά και ο καταναλωτής από την άλλη και δεν έχουν κανένα μέσο να αντιμετωπίσουν αυτή την αστάθεια αυτή τη στιγμή αυτοί οι δύο. Όλοι όμω αποδέχονται την αστάθεια όσο έχει αυτή τη στιγμή στο χρηματιστήριο και κανένα δεν κατανοεί ε, ακριβώς ε, το μέγεθο τη αστάθεια που αντιμετωπίζει ο ίδιο ο παραγωγό. Όλοι σκεφτόμαστε μόνο την αστάθεια στο χρηματιστήριο. Αυτό είναι κάτι που έχουμε ήδη δει τώρα. Η ε, κατηγορία 3 στο γάλα που χρησιμοποιείται και το τυρί. Βλέπετε την τιμή στον ιστορό ε, και κάτω την, το χρόνο από το 1980 μέχρι σήμερα. Με την μπλε γραμμή λένε οι Αμερικανοί ότι έχουν ελεύθερη αγορά, όμως έχουν και μια στήριξη ενίσχυση των τιμών που είναι αυτή η μπλε γραμμή. Ε, και στην κόκκινη γραμμή έχετε τις τιμές ε, του γάλακτος της τάξης 3. Μέχρι τις αρχές του 90 ήταν, συμπορεύονταν αυτές οι δύο γραμμές και ουσιαστικά η ενίσχυση των τιμών κρατούσε τους, παραγωγού, τους παραγωγούς που δεν ήταν βιώσιμοι στην αγορά. Συνέχισαν λοιπόν να παράγουν, δεν υπήρξε επίπτωση στην αγορά. Με... Έφτασαν όμως αυτές οι ενισχύσεις σε ένα επίπεδο που έπρεπε οι παραγωγοί να πάρουν την εμπορική απόφαση να βγουν από την παραγωγή και έτσι υπήρξε αύξηση της τιμής λόγω της πτώσης της παραγωγής. Δεν είναι μόνο αυτό βέβαια η αιτία, όμως το καλύπτει εν μέρη. Το ίδιο βλέπουμε και εδώ στην Ευρώπη, στην επόμενη διαφάνεια θα το δείτε. Η τιμή του βουτύρου λοιπόν, τα επίπεδα παρέμβασης έφτασαν σε τέτοιο βαθμό που πλέον δεν ήταν εμπορικά βιώσιμο για κάποιους παραγωγούς να παραμείνουν στην παραγωγή, βγήκαν από την παραγωγή, έπεσε η παραγωγή, αυξήθηκε η τιμή και έτσι μειώθηκε η τιμή. Το ίδιο βλέπουμε και στην επόμενη διαφάνεια βασικό σκοπός της διαχείρισης κινδύνου είναι η διαχείριση των ορίων, των περιθωρίων, να ε, περιοριστεί ε, η, αστάθεια και να διασφαλίσουμε τα έσοδα. Είναι δύσκολο να διαχειρίσουμε τους ε, κινδύνους με μία ανεξάρτητο τρόπο. Αφενός οι παραγωγοί προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι θα έχουν τις υψηλότερες δυνατές τιμές και από την άλλη ε, οι καταναλωτές θέλουν τις χαμηλότερες δυνατές τιμές. Πρέπει λοιπόν να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Πώς γίνεται αυτό. Επόμενη διαφάνεια. Πώς λειτουργεί τώρα αυτό το σύστημα στην Αμερική. Ε, τώρα, μέσω των ε, συνεταιρισμών, οι χρήστες από πλευράς παραγωγών παίρνουν την ίδια τιμή κάθε μήνα, τιμή μεταβλητής ή μπορούν εθελοντικά να πάνε στο συνεταιρισμό τους και να προσδιορίσουν, να καθορίσουν την τιμή. Εδώ είναι ένα γράφημα για τα επόμενα δύο χρόνια και έτσι μπορούν οι Αμερικανοί παραγωγοί να, τιμήσουν μια να πωλήσουν το γάλα τους σε μια προκαθορισμένη τιμή για τα επόμενα δύο χρόνια ή ένα ποσοστό του γαλακτός τους. Αυτό προσπαθούμε να ε, κάνουμε και εδώ στην Ευρώπη. Εδώ βλέπετε την τιμή του γάλακτος ε, της κατηγορίας 3 στην Αμερική. Ο Γιώργος λοιπόν παίρνει την τιμή με βάση αυτή την διαβαθμισμένη τιμή. Επομένως, η πράσινη γραμμή βλέπετε εδώ. Στο τέλος της κόκκινης γραμμής είναι εδώ που βρισκόμαστε τώρα το 2016, στην τιμή του γάλακτος. Πράσινη γραμμή, ο Γιώργος μπορεί να ε, πάρει τηλέφωνο το συνεταιρισμό και να πει ότι θέλω ε, ένα ε, ποσοστό του γάλακτός μου να απολυθεί σε αυτή την τιμή και να έχει λοιπόν ασφάλεια σε ό,τι, και διαβεβαίωση ότι αφορά εγγύηση τιμής για τα επόμενα δύο χρόνια για ένα ποσοστό ή για το σύνολο της παραγωγής γάλακτος. Αυτό είναι το πιο ε, σημαντικό γράφημα θεωρώ της παρουσίασης γιατί ξέρω ότι δεν έχω και πολύ χρόνο. Ε, γαλακτομική παραγωγή στην Αμερική, η κόκκινη γραμμή είναι η κατηγορία, η τιμή του γάλακτος κατηγορίας 3 που ισχύει για τους παραγωγούς στην Αμερική. Έχουν ένα πρόγραμμα κάλυψη κινδύνου για του γεωργού, για του παραγωγού. Βλέπουμε ότι έχουμε υψηλέ και χαμηλέ τιμέ στην κόκκινη γραμμή. Μπλε γραμμή είναι η μέση τιμή ε, για την οποία κάνουν κάλυψη κινδύνου οι παραγωγοί. Έτσι έρεται η ακραία αστάθεια. Έτσι δεν αποφελούνται των πολύ υψηλών τιμών, αλλά δεν πλήττονται και από τι πολύ χαμηλέ. Τελικά λοιπόν επιτρέπουμε στους παραγωγούς να προγραμματίσουν ε, και να σχεδιάσουν το μέλλον τους. Γιατί είναι μια επένδυση του αντίστοιχου 40 σέντε το λίτρο στην Ευρώπη. Όταν κάποιο παίρνει 40 cent το λίτρο, ε, θα δανειστεί ο παραγωγό, θα αγοράσει τρακτέρ και το καθεξή. Τι θα γίνει όμω μετά από μερικού μήνε που θα πέσει πάρα πολύ τιμή και δεν θα μπορεί να ε, αποπληρώσει το δάνειο στην τράπεζα. Έτσι, με, αυτή την κατάσταση βλέπετε ότι ε, στα, 30 σε το λίτρο μπορεί κάποιο να πάρει δάνειο και ξέρει ότι θα μπορεί να το αποπληρώσει τα επόμενα δύο χρόνια θα μπορούσε τώρα να λειτουργήσει αυτό στην Ευρώπη. Θα πέρασε κάποιε διαφάνειε. Εδώ βλέπετε πού θα μπορούσαν να είχαν καθορίσει την τιμή με την κάλυψη κινδύνου η παραγωγή. Το Μάιο του 2014. Ουσιαστικά ε, βλέπουμε την τιμή του γάλακτο για του παραγωγού. Αυτή τη στιγμή παίρνουν 30 cent το λίτρο. Το Μάιο του 2014 θα μπορούσαν να είχαν κλειδώσει μια τιμή με αυτά τα εργαλεία πάνω από τα 36 cent το λίτρο. Θα είχε λοιπόν δώσει δυνατότητα την πρόσβαση ε, των παραγωγών στην αγορά και ε, μια ασφάλεια. Θα μπορούσε λοιπόν να έχει κλειδώσει την τιμή ο παραγωγό σε μια υψηλότερη κατά 5,6 cent καλύτερα τιμή. Και αυτό θα έχει προστατεύσει και το περιθώριο κέρδους του. Συγγνώμη που τρέχω, επόμενη διαφάνεια. Εδώ έχετε το ισοδύναμο για έναν Βρετανό παραγωγό. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή παίρνουν 15-20 ε, λεπτά της ε, λίρας. Ε, θα ήταν υψηλότερο αν το είχαν κάνει πιο νωρίς. Κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχει ρευστότητα στην αγορά. Αυτό δεν ισχύει ουσιαστικά. Καθημερινά κλειδώνουμε χιλιάδες τόνους προϊόντος για ορισμένες οικονομικές, οικονομικούς φορείς προχάραμε στο τέλο. Και συγγνώμη που υπερεύει το χρονικό όριο. Σα ευχαριστώ κύριο Σκάρλ για 8 λεπτά. Euh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτη διαφάνεια. και να απαντήσω στην ερώτηση που υποβάλλατε προηγουμένως για τα αίτια της αστάθειας των τιμών. Μεταξύ των αιτίων βρίσκονται και οι προσδοκίες των γεωργών, οι κερδοσκοπίες και οι φυσικοί κίνδυνοι. Οι πρώτοι δύο κίνδυνοι είναι εξωγενείς, δηλαδή δεν εξαρτώνται από τους, ε, εξαρτώνται από τους ίδιους τους ε, συντελεστές και άρα δεν είναι ασφαλιστέοι οι μόνοι κίνδυνοι που μπορούν να τύχουν ασφάλισης είναι οι κλιματικοί, καιρικοί παράγοντες. Και αυτό καθορίζει την αστάθεια των τιμών και τη φύση των κινδύνων που έχουμε να διαχειριστούμε. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Η αστάθεια των αγορών είναι διαρθρωτική και η κατάργηση των δημόσιων πολιτικών και κυρίως της αποθεματοποίησης ε, οδήγησε σε μια αστάθεια που ε, είναι σήμερα πιο δύσκολο να τη διαχειριστούμε. Ε, παλιά μπορούσαμε να το κάνουμε με την αποθεματοποίηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να επανέλθουμε στην αποθεματοποίηση, αλλά η αποθεματοποίηση πρέπει να είναι το μέτρο, αλλά να υπάρχει και καλό θα είναι να το έχουμε αυτό κατά νου. Ε, τι γίνεται με την αστάθεια. Όταν έχουμε ε, μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης και έχουμε ε, κάποια αποτελέσματα όμως που ε, ξεπερνούν τις διαφορές μεταξύ προσφοράς και της ζήτησης και πλήττουν το σύνολο της οικονομίας. Εδώ, όπως είπε ο κύριος Φέντον, έχουμε για την αγορά γάλακτος τα τελευταία δέκα χρόνια τεράστιες διακοιμάσεις, όλο και πιο μεγάλες ε, και ακραίες. Έχουμε διπλάσεις, τετραπλάσεις διακοιμάσεις από τις συνηθισμένες ε, και έχουμε διαφορές 10% ετησίως, τεράστια ποσά και ίδιες διαφορές ισχύουν και για τα σιτηρά, για το σιτάρι. Από τις αρχές του 2000 είχαμε αστάθειες ε, όλο και μεγαλύτερες στις τιμές και όλο και μεγαλύτερες διακοιμάνσεις. Μπορεί να έχουμε ε, περίοδες χρόνων αγελάδων που μπορεί να κρατήσουν ένα ή δύο χρόνια, κανένας όμως δεν μπορεί να το προβλέψει. Επίσης, τα οικονομικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για να στηρίξουν τις πολιτικές αποφάσεις, το μοντέλο της Παγκόσμιας Τράπεζας ή του ΟΣΑ, κατά τη γνώμη μου, έχουν κάποια προβλήματα στην πρόβλεψη της αστάθειας, γιατί θεωρούν ότι η προσφορά προσαρμόζεται αυτόματα στις τιμέ. όλοι οι συντελεστέ έχουν εύλογε προσδοκίε, κάτι που δεν ισχύει, δεν λαμβάνονται υπόψη καιρικέ συνθήκες και περιβαλλοντικοί παράγοντες, επίσης ε, το, ο ρόλος των αποθεμάτων και δεν λαμβάνεται υπόψη και ο ρόλος των κερδοσκόπων. Επίσης έχουμε τις προβλέψεις ε, του μοντέλου του ΟΣΑ για κάθε χρόνο από το 1990. Οι προβλέψεις ε, είναι αυτές που γίνονται κάθε χρόνο για τις εξελίξεις των τιμών συντηρών στη μαύρη γραμμή έχουμε την πραγματική εξέλιξη των τιμών. Καμία ορατότητα και καμία δυνατότητα πρόβλεψης της αστάθειας. Οπότε οι πολιτικοί ηθήνοντες καταργούν τις, τους μηχανισμούς παρέμβασης γιατί όταν το βλέπουμε αυτό νομίζουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα σταθερό περιβάλλον χωρίς κινδύνους, κάτι που δεν ισχύει. Επίσης, το μοντέλο της Μόμαγκρη, μας, ε, του δικού μας επιστημονικού επιτελείου, για να διαχειριστούμε αυτή την αστάθεια των τιμών. Βλέπετε τέλη του 2014 και την αναμενόμενη αστάθεια στις τιμές ετηρών μεταξύ του 2015 και του 2022. Βλέπετε ότι προβλέψαμε την μεγάλη μείωση του 2015 που συνεχίζεται το 2016. Θα έχουμε όμως πολύ σημαντικές διακυμάνσεις και δεν βρισκόμαστε σε ένα σταθερό περιβάλλον ή σταθεροποιημένο. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε ένα όργανο, ένα μηχανισμό για να προβλέψουμε αυτές τις αστάθειες. Επίσης, ποια είναι τα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την ε, μεταβλητότητα, ε, την αστάθεια, τις φοβερές διακοιμάσεις. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι δεν υπάρχει πανάκια, δεν υπάρχει θαυματουργή λύση. Και στις ερωτήσεις που ακούσαμε, ε, διαπιστώνουμε ότι οι ευρωβουλευτές προσπαθούν να βρουν κάποιες προβλέψεις για την εξέλιξη της ΠΑΚ. Δεν υπάρχει προβλέψιμη μεταρρύθμιση. Για παράδειγμα, αποθεματοποίηση, εποχικότητα, εναλλακτικές, ε, εναλλακτικές διέξοδοι, τα βιοκαύσιμα. Καλύτερα πρόληψη σίγουρα παρά θεραπεία. Είναι λιγότερο δαπανηρή η πρόληψη. Επίσης, ποιες είναι οι δυνατές, ποιοι είναι οι δυνατοί μηχανισμοί παρέμβασης. Καταρχήν, έχουμε τους μεμονωμένους ή τους συστημικούς κινδύνους. Έχουμε επίσης ε, καταστροφικούς κινδύνους ή ελέγξιμους κινδύνους. Είναι προφανές ότι η δημόσια παρέμβαση θα πρέπει να βρίσκεται ψηλά δεξιά για να μπορέσει να ε, επανισορροπήσει τις αγορές με αντικυκλικές ενισχύσεις και ε, αλληλεγγύη για τις θεομηνίες, γιατί έχουμε ταυτόχρονα και καταστροφικούς και συστημικούς κινδύνους. Αυτό βλέπουμε στον τομέα του γάλακτος αυτή τη στιγμή και σε μερικούς τομείς της κτηνοτροφίας. Σε ό,τι αφορά τους ελέγξιμους κινδύνους, εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε πιο ε, συλλογική παρέμβαση και πιο συνεργατική, όπως είπε ο κ. Φέντον, και να αξιοποιήσουμε την, ανάγκη, το, την δυνατότητα των συνεταιρισμών ή των κλάδων να μετριάσουν την αστάθεια και να επηρεάσουν το ύψος των τιμών. Επίσης έχουμε κάποια ταμεία επιμερισμού των κινδύνων ή προθεσμιακές καλύψεις ή ασφάλειες των ε, εσοδιών από τους κλιματικούς κινδύνους. Επίσης, θα πρέπει να βρούμε τους μηχανισμούς παρέμβασης. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνουν σε εθνικό επίπεδο. Είτε σε ασφάλεια εισοδήματος, είτε στον επιμερισμό των κινδύνων. Ε, το κοινωτικό σύστημα προβλέπει ε, είτε ελαστικότητα στα κράτη-μέλη διακριτική ευχέρεια, είτε ε, βοήθεια από το κοινοτικό προϋπολογισμό. Σε ό,τι αφορά τον ατομικό κίνδυνο, αυτός ο κίνδυνος θα πρέπει να ε, τύχει διαχείρισης σε επίπεδο εκμετάλλευσης, ενώ ο συστημικός κίνδυνος θα αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο. Με την εξισορρόπηση, με την μείωση των βαρών για παράδειγμα, το διαπιστώσαμε αυτό στη Γαλλία και πουθενά στο πίνακα αυτό διαχείριση των κινδύνων δεν βρίσκουμε τι αποσυνδεδεμένε ενισχύσει. Γιατί οι αποσυνδεδεμένε ενισχύσει δεν επηρεάζουν καθόλου τη διαχείριση τη αστάθεια και τη διαχείριση των κινδύνων. Και γνωρίζουμε ότι το 60% του ευρωπαϊκού προπολογισμού αφιερώνεται στι αποσυνδεδεμένε ενισχύσει, που είναι άχρηστε για να αντιμετωπίσουμε την αστάθεια των τιμών, είτε προ τα πάνω είτε προ τα κάτω. Και επίσης καλό θα ήταν ε, να, γίνει μια ανακατανομή των αποσυνδεδεμένων ενισχύσεων προς τις αντικυκλικές ενισχύσεις για να επανισορροπήσουμε τις αγοράς. Και στο σχέδιο μεταρρύθμισης της ΚΑΠ που εκπονούμε διαπιστώνουμε ότι θα, ε, θα μας κόσει πολύ λιγότερο ένα τέτοιο σύστημα ε, και σε περίοδο ισχνών και σε περίοδο παχιών αγελάδων. Επίσης για την περίοδο 2011-2015 θα είχαμε εξοικονομήσει 7 με 8 δισεκατομμύρια το χρόνο και σε περίοδο κρίση όπως η σημερινή το κόστος θα ήταν αντίστοιχο με το κόστος του που προβλέπεται στις πολιτικές ε, προοπτικές, στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Οπότε με αντικυκλικά μέτρα ή με μέτρα παρέμβαση των αγορών θα είχαμε πολύ, πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι με το σημερινό σύστημα γιατί σήμερα αφιερώνουμε πολλά κονδύλια σε ενισχύσεις που δεν επηρεάζουν καθόλου ούτε τη διαχείριση των κινδύνων, ούτε τη διαχείριση της αστάθειας των τιμών. Σε έναν ανοιχτό αποκοσμιοποιημένο κόσμο θα πρέπει οπωσδήποτε να προσαρμόσουμε την κοινή γεωργική μας πολιτική. Ευχαριστώ. Μάλιστα, μας δώσετε τροφή για σκέψη. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους ε, προηγούμενους μας εμπειρογνώμονες για σύντομο σχολιασμό. Πρώτα στον κύριο Φερέρ για δύο λεπτά. Αυτό που διαπιστώνουμε και είμαι υποχρεωμένος να το επαναλάβω είναι να διαπιστώσουμε αν, είναι να εξακριβώσουμε αν θα εμείνει η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση στη διαχείριση της κρίσης ε, προσπαθώντας να ε, κάνει μια πρόοδο γιατί το 2003 ε, ελήφθη απόφαση για την αποσύνδεση ώστε να είμαστε σε καλύτερη διαπραγματευτική θέση για την Τόχα. Δεν έχουμε καταλήξει το γύρο της Τόχας, αλλά ήδη έχουμε μετα... ε, υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις. Είναι πολιτικό θέμα. Επίσης, η πραγματικότητα της αστάθειας των τιμών. Η αστάθεια των τιμών ε, οδήγησε την Γεωργία ε, στην εποχή του Φαραώ. Δηλαδή έχουμε περιόδους παχιών και ισχνών αγελάδων. Οπότε έχουμε σίγουρα τρία μέτρα πρόληψης ή διαχείρισης που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε. Καταρχήν, ε, μέτρα εξασφάλισης ε, απέναντι στην αστάθεια. Θα πρέπει να διδάξουμε ή να ξαναμάθουν οι γεωργοί και οι ε, οργανώσεις παραγωγών πώς θα διαχειριστούν τις περιόδους ισχνών και παχιών αγελάδων. Όταν έχουμε περίοδο ακμής να βάζουν κάτι στην άκρη για να μπορέσουν ε, στις ε, περιόδους παρακμής να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια μέτρα σταθεροποίησης, αλλά σίγουρα θα πρέπει να στηρίζονται στην κατάρτιση αλλά και σε φορολογικά μέτρα εθνικά και ε, κοινοτικά. Επίσης, ε, η διαφοροποίηση, να επενδύσουμε στη διαφοροποίηση της παραγωγής. Όσο περισσότερες μονοκαλλιέργειες έχουμε, τόσο πιο ευάλωτοι θα είμαστε στην αστάθεια των τιμών. Θα πρέπει να καλλιεργήσουμε διαφοροποιημένη, μια ανατροπία διαφοροποίησης ε, της γεωργίας να μην βάζουμε όλα τα αυγά μας στο ίδιο καλάθι. Επίσης, μέτρα ασφάλισης και μέτρα πιο αποτελεσματική στήριξη. γιατί έχουμε ξεπεράσει τα όρια μας. Θα πρέπει οι δημόσιες αρχέ τώρα να στηρίξουν τους γεωργούς, ώστε η ανθεκτικότητά τους ε, να ενισχυθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σαντινόλφη. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο και εκ μέρου μου. Ε, προφανώς το θέμα των χρηματοπιστωτικών αγορών είναι ένα στοιχείο κάλυψης ε, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσω και εγώ κάτι ε, σε σχέση με αυτά που ελέγχθησαν για την αστάθεια των τιμών. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά στοιχεία που παίζουν ρόλο και άλλα πάλι όχι. Θέλω όμως να πω το εξής, ότι οι χρηματοψηφιακές αγορές δεν καλύψουν όλες τις ε, γεωργικές ε, παραγωγές. Άρα δηλαδή ε, θα πρέπει να εισαχθεί και στη γεωργική παραγωγή αυτό το στοιχείο της κάλυψης. Ανάλογα βέβαια και με το είδος της παραγωγής και της καλλιέργειας. Υπάρχει ένα σημαντικό θέμα, το θέμα της διαχείρισης των κινδύνων. Αυτά είναι καθοριστικά στοιχεία που μας ε, επιτρέπουν να κατανοήσουμε ποιος πρέπει να παρέμβει και πού. Πιστεύω λοιπόν ότι από τη στιγμή που θα υπάρχει διαφάνεια και από τη στιγμή που θα υπάρχει ε, συνεργασία, αυτά είναι στοιχεία ε, που έχουν επικρατήσει στην Ευρώπη. Δηλαδή, η αγορά να είναι μόνο πιο διαφανής, αλλά πρέπει να υπάρχουν και κάποια στοιχεία που θα βοηθούν να μπορεί κανείς ε, να παρέμβει όταν οι ε, εποχές, όταν οι αγορές είναι καλές και όταν υπάρχει ακόμα και κρίση. Δεν υπάρχει μία ενιαία λύση για να προστατευτούν οι γεωργοί από τα διάφορα από τους κινδύνους. Βεβαίως μπορούν να υπάρχουν συμπληρωματικές καλύψεις. Αυτό το Ταμείο Αμοιβαιοποίησης θα μπορούσε να είναι ε, μια στρατηγική, αλλά είναι ένα πολύ περίπλοκο ε, στοιχείο της συζήτησης. Εγώ πάντως ε, θέλω να πω ότι όσον αφορά τη συζήτηση της αντικυκλικότητας, θέλω να σας πω ότι οι άμεσες πληρωμές στην Ευρώπη δεν είναι ο μόνος μηχανισμός ε, και δεν είναι μόνο μηχανισμός στήριξης ε, του εισοδήματος. Εμείς λοιπόν κάνουμε όλες αυτές τις σκέψεις ε, βεβαίως για να δούμε κατά πόσον θα μπορούσε να υπάρχει στο μέλλον ένα σύστημα που θα επιτρέπει μια τέτοια φιλοσοφική προσέγγιση έτσι ώστε οι άμεσες πληρωμές να είναι ένα είδος στήριξη του εισοδήματος. Ευχαριστώ. Και τώρα ο λόγος των εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον κύριο Χανιώτη. Παρακαλώ κύριε Διευθυντά, έχετε το λόγο. Ο uh, moment. Συγγνώμη. Πρέπει πρώτα να δώσω το λόγο στον τρίτο μας εμπειρογνώμονα, στον κύριο Μπέιση για το σχολιασμό, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Χανιώτη. Νομίζω ότι αυτά που είπαν οι συνάδελφοί μου είναι πολύ ενδιαφέρουσες ε, απόψεις σχετικά με την αστάθεια των τιμών, αλλά όπως ήδη διαπιστώθηκε δεν υπάρχει μία μαγική συνταγή ε, σε σχέση με αυτά που πήρε ο κύριος Φαντόμ, δηλαδή η κάλυψη των αγορών. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο δεν είναι πολύ συναντισμένο στην γαλακτοκομική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τουλάχιστον γνωρίζουμε ότι οι γεωργοί που χρησιμοποιούν χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία επιθυμούν να έχουν περαιτέρω στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορούν να προστατεύονται και από χαμηλέ τιμέ. Και βλέπουμε το ίδιο και στι Ηνωμένε Πολιτείε, όπου το σύστημα υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, είναι αρκετά διαδεδομένο. Όμω οι γεωργοί παρόλα αυτά βασίζονται ε, σε αυτό που αναφέρθηκε ήδη, δηλαδή στο πρόγραμμα προστασία του περιθωρίου στα γαλακτοκομικά. Δεν λέω ότι είναι κάτι που δεν λαμβάνεται υπόψη, αλλά από την άλλη, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει περαιτέρω περιθώριο για τις κυβερνήσεις για να μπορούν να παρέμβουν. Ακούστηκε η ιδέα των ε, άμεσων πληρωμών να είναι αντικυκλικές. Καλό αυτό να το εξετάσουμε περαιτέρω, παρότι θέλω να πω εδώ πρέπει να είναι σαφές ότι αυτό δεν πρέπει να συνδέεται με την παραγωγή, γιατί αν συμβεί κάτι τέτοιο δεν θα έχουμε επαρκή εφαρμογή, ικανοποιητική εφαρμογή, αντικυκλικές ε, πληρωμές που δεν συνδέονται με την παραγωγή, συνδέονται όμως με ε, περιβαλλοντικές ε, προϋποθέσεις, στις ΗΠΑ υπήρξε μια τέτοια ιδέα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας για τον πρώτο πινόλα στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτικής. Προφανώς δεν έχω κι εγώ μια σαφή λύση για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν όλα αυτά. Θα εξαρτηθεί βέβαια από τα κράτη-μέλη αλλά και από κάθε συγκεκριμένα τομέα γιατί τα πράγματα ποικίλουν. Εξάλλου πρέπει να εξετάσουμε με λεπτομέρειες το πώς ακριβώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στο να κερδοσκοπούν οι γεωργοί στις, σε σχέση με τις ε, καταβαλλόμενες ενισχύσεις. Αυτό συμβαίνει κυρίως στις ΗΠΑ. Πολιτείες. Άρα δηλαδή οι πληρωμές που καταβάλλονται στους γεωργούς δεν κεφαλοποιούνται σε άλλες μορφές όπως συμβαίνει κατά πάσα πιθανότητα με τις άμεσες πληρωμές. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ήρθε η σειρά του κύριου Χανιώτη. Παρακαλώ κύριε Διευθυντά, έχετε το λόγο. Thank you very much, uh, for us the... Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που μας δίνει τη δυνατότητα να σχολιάσουμε ορισμένα ε, στοιχεία αυτή της ακρόασης. Ε, θα σταθώ και στα τρία σημεία που έχετε θέσει στην ημέρα διάταξη. Σαφώ και η αστάθεια δεν αφορά μόνο τις γεωργικές αγορές... Ε, συνδέεται με το γεγονό ότι η ζήτηση είναι συνεχής και καθημερινή, ενώ η προσφορά ε, δεν είναι τόσο συνεχής, εξαρτάται και από την ε, προτεραιότητα της παραγωγής και από τον καιρό τον ίδιο και γι' αυτό δεν κατανοώ και τη σύνδεση με την ηλεκτρική ενέργεια γιατί πρέπει να είναι συνεχής η προσφορά, δεν υπάρχει αγορά. Το πιο πρόσφατο ενδιαφέρον για τον αντίκτυπο της αυστάθειας των τιμών στην γεωργία και στα τρόφιμα ε, κατευθύνεται από αυτό που θεωρείται γενικά ως ε, υπερβολική αστάθεια των τιμών και τις ε, δυσκολίες που ε, δημιουργεί από το σχεδιασμό της παραγωγής μέχρι και τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Στην Γενική Διάθεση εμείς αναλύουμε τις εξελίξεις αυτές από την άξη των τιμών του 2008 και το συμπέρασμά μας είναι ότι το πιο ανησυχητικό δεν είναι η αστάθεια ε, που δεν αυξήθηκε καθόλου μάλιστα σε όλα τα προϊόντα ε, και καθόλου τη διάρκεια μετά το 2008. Παράλληλα, μάλιστα, θεωρούμε ότι η ε, συνύπαρξη τριών παράλληλων τάσεων είναι το ενισχυτικό. Η αστάθεια, η κίνηση, παράλληλη κίνηση όλων των τιμών των εμπορευμάτων και η για τα μελλοντικά επίπεδα τιμών. Η συμφωνία του ΠΟΕ υπογράφηκε το 1995, ενώ οι μεγάλες ε, αυξήσεις τιμών παρατηρήθηκαν το 2004. Δεν έχουν σχέση με τον ΠΟΕ, έχουν σχέση με τις μακροοικονομικές εξελίξεις που οδήγησαν ε, στην κρίση του 2008. Ιδίω τα επίπεδα των τιμών, παρότι είναι πιο υψηλά από τα ιστορικά υψηλά, ε, μετά από την μια αντιστροφή της καθοδικής πορείας στο παρελθόν, είναι η πηγή της μεγαλύτερης ανησυχίας. Κατά τη γνώμη μας, ιδίως αν δείτε ε, τάσει των τιμών σε συγκεκριμένε περιόδου, βλέπουμε ότι η μεγαλύτερη ανησυχία των γεωργών συνδέεται με το γεγονό ότι μέσα σε 8 χρόνια έχουν δει δύο φορέ τι τιμέ να φτάνουν σε δυσθεώρητα ύψη ε, και να πέφτουν ε, σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Αν δείτε λοιπόν ε, το κάτω μέρος, όπου έχουμε την περίοδο 97-2015, ε, ξεκινήσαμε από την προηγούμενη μεγάλη αύξηση των γεωργικών εμπορευμάτων οι γεωργικέ τιμέ σε πραγματικούς όρου είναι 10% υψηλότερε σε σχέση με πριν από 10 ε, χρόνια. Τα λοιπάσματα 100%, τιμέ ενέργεια 95% και βεβαίως ε, μεταλλεύματα και ορυκτά επίσης ε, υψηλότερε τιμές. Έχουμε λοιπόν επιδείνωση και αυτή η επιδείνωση είναι το, το, το αντικείμενο εδώ. Ε, οι γεωργικές τιμές ε, βρέθηκαν στο επίκεντρο της καθοδικής ε, τάσης ε, μέσω εξελίξεων λόγω της επιβράδυνσης της οικονομίας και στην Κίνα και σε άλλες αναδυόμενες οικονομίες και ε, προκαλείται από την υπερβολική, από την υπερπροσφορά και αυτό ισχύει και για το φυσικό αέριο. Η μεγάλη προσφορά που προκύπτει από τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και την υπερβολική αντίδραση στο προηγούμενο ευνοϊκό περιβάλλον επίσης αποτελούν σημαντικό τμήμα της καθοδικής ε, τάσης. Και το ρωσικό εμπάργκο βεβαίω δεν έχει βοηθήσει, ιδίω στα γαλακτοκομικά. Όμω βλέπουμε το ενδιαφέρον ότι αυτή η πρόσφατη καθοδική ε, τάση δεν χαρακτηρίζεται από την αύξηση στην αστάθεια, Όπω δείτε στην επόμενη διαφάνεια. Αν δείτε τις αιτήσιες ε, μεταβολές ε, στι πραγματικέ τιμέ, σε παγκόσμιο επίπεδο, βλέπουμε ότι υπάρχει η τάση της αστάθειας, αλλά λιγότερο από ό,τι στο παρελθόν. Στα λοιπάσματα είναι πολύ υψηλότερη και στην ενέργεια. Το σημαντικό είναι αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια έχουμε μια παράλληλη ε, καθοδική τάση στις τιμές. Και αν δούμε τα μηνιαία στοιχεία των τιμών ε, σε, σε ονομαστικούς όρους και πάλι η μηνιαία μεταβολή των γεωργικών τιμών, βλέπετε τι συμβαίνει και στα λοιπάσματα και στην ενέργεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη αστάθεια σε κάποια πορεύματα, σε κάποια προϊόντα από ό,τι σε άλλα. Ούτε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένε ε, περίοδοι όπου είχαμε αύξηση τη αστάθεια. Όμω σημαίνει ότι αν δούμε γενικότερα, τη γενικότερη εικόνα, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα από ό,τι νομίζουμε. Τα ξέρετε τα μέτρα τη κοινή γεωργική πολιτική, δεν ήρθα εδώ να σα τα εξηγήσω και πάλι. Ήθελα μόνο να επισημάνω ε, σε αυτό το γνωστό διάγραμμα ε, για την εξέλιξη της ΚΑΠ, το μπλε κομμάτι είναι οι συνδεδεμένε ενισχύσει. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της ε, συμφωνίας ε, ΠΟΕ. Η συνδεδεμένη ενίσχυση ήταν ε, αποτέλεσμα της προετοιμασία για τη διεύρυνση και για την κρίση με, ε, με την ασθένεια των τρελών αγελάδων. Και έπρεπε να έχουμε μεγαλύτερο προσανατολισμό με την αγορά προς την αγορά στους παραγωγούς. Βλέπετε εδώ πέρα την γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των τιμών Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκόσμιας αγοράς. Και βλέπετε στο μπλε ε, τις τιμές στα γαλακτοκομικά το 2010 ότι ήταν ήδη σε επίπεδα παγκόσμιας αγοράς, όχι τον περασμένο Απρίλιο. Το ίδιο ισχύει και στα Δημητριακά, όπου η μεταρρύθμιση έλαβε χώρα πολύ πιο παλιά. Δεν έχουμε φτάσει σε επιθυμητό σημείο στη ζάχαρη και ε, στο βόλιο κρέας. Και ε, βεβαίως αυτό συνδέεται και με ωφέλη, όπως βλέπετε ε, στην επόμενη διαφάνεια, που είναι η θετική εξέλιξη των ε, γεωργικών συναλλαγών και των τροφίμων που συνδέονται με τη γεωργία, το οποίο έχουμε σπάσει σε διάφορες κατηγορίες, γιατί δεν είναι μόνο τα εμφιαλωμένα που έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές, είναι ένα ευρύ φάσμα προϊόντων. Εδώ υπήρξε μια φορά στην αντιμετώπιση επιμέρους ε, κατηγοριών κινδύνου. Οι κίνδυνοι της αγοράς που συνδέονται με εσωτερικές και εξωτερικές διαστάσεις της ενίας αγοράς και ευρύτεροι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, κίνδυνοι που συνδέονται συγκεκριμένα με τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών και, ή και των περιφερειών τους, ας πούμε, κίνδυνοι που συνδέονται με τον καιρό, με ασθένειες και γενικότερα φυσικά φαινόμενα και αβεβαιότητε ε, αντιμετωπίζονται σε επίπεδο κράτου μέλου. Όμω κάτι το οποίο παραγνωρίζουμε ή κάτι που διαστρεβλώνεται συχνά στην συζήτηση είναι ο αντίκτυπο των πλέον στοχοθετημένων μέτρων πολιτική που ε, στόχο έχουν την αντιμετώπιση ακριβώ τη αστάθεια των εισοδημάτων ή αποσυνδεδεμένε άμεσε ενισχύσει. Στην πράξη αυτέ οι πληρωμέ διασφαλίζουν ένα ε, ευρωπαϊκό ε, σύστημα βασική στήριξη εισοδήματο που είναι ανεξάρτητο από τι ε, μεταβολέ τη αγορά, μειώνει, περιορίζει την αστάθεια των εισοδημάτων και διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση τη γεωργική ανταστηριότητας σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια και επιτρέπει την υποβοήθηση των παραγωγών για να αποφασίσουν οι ίδιοι πώς θα προσανατολιστούν στο μέλλον τις αποφάσεις τους δηλαδή. Τώρα η μεταβολή στην κοινή γεωρική πολιτική αντικατόπτρισε μια ε, επιλογή πολιτικής ως μια ανταπόκριση σε μια μακροπρόθεσμο, ένα μακροπρόθεσμο δίλημα στον φορά την γεωρική πολιτική. Τι είναι το καλύτερο ε, στην πράξη, η ε, η στοχοθέτηση των τιμών ουσιαστικά αυξάνει τις τιμές γιατί δίνει κίνητρα για την υπερβολική παραγωγή το οποίο τελικά οδηγεί σε περαιτέρω πτώση των τιμών και τελικά έχουμε έναν φαύλο κύκλο. Αυτό μπορεί να, αυτή η συνταγή μπορεί να λειτουργήσει προσωρινά για μικρές ή απομονωμένες χώρες, όμως δεν σταθεροποιεί τα εισοδήματα στις ανοιχτές οικονομίες συχνά έρχομαι στην αντιμετώπιση με το ζήτημα για το αν και κατά πόσο η αμερικανική προσέγγιση ε, είναι κατάλληλη για την κοινή γεωργική πολιτική, το οποίο ανέκυψε και σήμερα. Είναι πολύ σημαντική και η γεωργική ε, πολιτική της Αμερικής και η Αμερικανική γεωργία για το παγκόσμιο εμπόδιο, ε, εμπόριο. Συγνώμη. Όμως πρέπει να έχουμε κατά νου τις θεσμικές, δημοσιονομικές και διαφορετικές διαφορές μεταξύ των δύο εταίρων. Δεν υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί στην υλοποίηση της αμερικανικής πολιτικής και η αμερικανική πολιτική βασίζεται στην ε, ε, προσφορά ε, σε μία σε τεράστιες γεωργικές εκτάσεις και στην πρωτογενή χίδιν παραγωγή προϊόντων. Επομένω, δεν πρέπει να τα υπεραπλουστεύουμε τα πράγματα. Όπω και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αμερικανικέ πολιτικέ είναι συμπληρωματικέ η μία προ την άλλη και αντικατοπτρίζουν πολύ διαφορετική φιλοσοφία από αυτή που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, κατά πόσο πρόκειται για αντικυκλική στήριξη των τιμών ή ε, καθεστώτα ε, ασφάλιση, όπω και να έχει, οι αμερικανικέ πολιτικέ επιτρέπουν σε ένα τμήμα τη αμερικανική γεωργία να απομονωθεί από τα υπόλοιπα. Ε, μάλλον βραχυπρόθεσμα. Ε, βλέπουμε ότι το 60% των αμερικανικών πληρωμών πηγαίνουν σε ε, καθεστώτα διαχείριση κινδύνου και πάνω από 90% ε, αφορούν μόνο συγκεκριμένες καλλιέργειες όπως είναι ο αραβόστος και η σόγια για παράδειγμα. Όμως βλέπουμε και αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα και αν συγκρίνουμε τα αποτελέσματα την τελευταία δεκαετία είναι σαφή η εικόνα τα ευρωπαϊκά εισοδήματα γεωργικά είχαν μικρότερη αστάθεια και έχουν πέσει πολύ λιγότερο από ότι τα αμερικανικά εισοδήματα των γεωργών τα, πρόσφατα χρόνια, τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ 13 και 15 μάλιστα, 2013-2015, η πτώση του, του επιχειρηματικού εισοδήματο και του καθαρού εισοδήματο ήταν 6 και 14%, ενώ στην Αμερική ήταν 16 και 34%. Μεταξύ άλλων παραγόντων είναι και το αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η αναπόφευκτη προσαρμογή στην πραγματικότητα της αγοράς έρχεται πιο μετά και είναι πιο σημαντική στην Αμερικανική γεωργία παρότι στην ε, ε, Ευρωπαϊκή. Γιατί η Ευρωπαϊκή με το να μοιράζεται στήριξη σε όλο τον γεωργικό κλάδο επιτρέπει αλλαγές μεταξύ κλάδων και προϊόντων για να εξομαλύνουμε την ε, αστάθεια και την προσαρμογή σε αυτήν. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε μία τέτοια εξήγηση γιατί συγκρίνουν ε, την ανταπόκριση σε τιμή, σε χαμηλότερη ε, τιμή με τον αντίκτυπο μιας αντικυκλικής στήριξης. Όμως η αντικυκλική στήριξη δεν λέει στον παραγωγό τι τους δίνει η αγορά, τους λέει τι πληρώνει η κυβέρνηση που είναι η, η τιμή στόχος. Συμπερασματικά, πρέπει πρώτα να προσδιορίσουμε το πρόβλημα το οποίο θέλουμε να λύσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά να αποφασίσουμε τι άλλο θέλουμε να κάνουμε. Το Είναι το πρόβλημα το ότι το πρόβλημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η αστάθεια των τιμών και έτσι πρέπει να, να επικεντρωθούμε πιο πολύ στα προϊόντα. Εμεί θεωρούμε πω όχι. Πιστεύουμε ότι σε ό,τι αφορά και τα δημόσια και τα ιδιωτικά αγαθά, η αντιμετώπιση τη αστάθεια των εισοδημάτων θα πρέπει να είναι Βασικό στόχο και βασική πρόκληση, πρόκληση της κοινή γεωργική πολιτική. Και πολλά διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από την υλοποίηση των νέων εργαλείων και την έλλειψη ελκυστικότητα αυτών των ε, ε, εργαλείων, ότι δεν είναι πολύ δημοφιλή. Ε, αντίστοιχα και από το αμερικανικό, ε, σε ό,τι αφορά το όριο, περιθώριο για το γάλα, το οποίο επεκτάθηκε χρονικά δύο φορές, γιατί και πάλι δεν, υπήρχε, δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και περνάμε στη συζήτηση. Ζήτησαν το λόγο οι κύριοι Ντες, Ντόρφμαν, Ταραμπέλα. Άλλος κανείς για να δω πόσο χρόνο έχουμε και να τον κατανείμω μεταξύ των ομιλητών. Ροπέ. Πέντε λοιπόν συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Παρακαλώ χρόνου φίδου. Ο κύριος Ντες. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω να κάνω κάποιες προσθήκες. Πολύ σωστά ελέγχθη ότι δεν υπάρχει μαγική λύση. Τόντι στην Ευρώπη τα πράγματα ποικίλουν. Όμως έχω μία ερώτηση για το θέμα του καθορισμού των τιμών. Η τιμή του γάλακτος είναι στα 36 σέντ και αναφέρθηκε ήδη ότι για τα επόμενα χρόνια ε, υπάρχει μια συμφωνία να προσφέρεται το γάλα σε 32 cent. Όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει και ο συνεταιρισμό ε, να αγοράζει με χαμηλότερη τιμή γιατί αν ο συνεταιρισμό αγοράζει με 32 cent δεν θα μπορέσει να κρατήσει αυτή την τιμή και θα ήθελα να έχω μία απάντηση Πώς λειτουργεί αυτό. Επίσης κάτι άλλο που ελέγχθη, τα μεγαλύτερα προβλήματα τα έχουν οι νέοι γεωργοί οι οποίοι έχουν επενδύσει. Εδώ λοιπόν χρειαζόμαστε ένα σύστημα δανειοδότησης και πάω πάλι στο γάλα. 30 σέντ είναι το, το, το, ε, και ε, ανάλογα με το πόσο αυξάνεται η τιμή του γάλακτος, από εκεί εξαρτάται και το τοκοχρεολύσιο. Αν ε, δηλαδή ε, πέσει η τιμή του γάλακτος στα 10 cent, τότε δεν θα χρειαστεί να καταβληθεί κανένα τοκοχρεωλήσιο. Και η τελευταία μου παρατήρηση, στην Ευρώπη δεν είμαστε αρμόδιοι για τον κοινωνικό τομέα, όμως μπορώ να φανταστώ ότι θα βοηθούσε τους γεωργούς ε, ε, που καταβάλουν τις εισφορές τους ε, ασφάλειας ταινίας ε, συνταξιοδότησης να αναλαμβάνει το κράτος το 50% αυτό δεν θα είχε καμία επιρροή στις τιμές και θα ωφελούσε περισσότερο εκείνους οι οποίοι καλλιεργούν με την τεχνολογία μια μεγάλη έκταση πολλών εκταρίων. Θα ήθελα παρακαλώ να σχολιάσετε αυτό το οποίο είπα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην μιλάμε μόνο για την αστάθεια των τιμών, αλλά να μιλάμε κυρίως για την αστάθεια του εισοδήματος. Για τη τελική ανάλυση αυτό ενδιαφέρει τον Γεωργό και τον κτηνοτρόφο. Και κυρίως αν δει κανείς το γαλακτοκομικό τομέα, αν δει τους αριθμούς. Ε, το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό ε, στο γερμανικό, α, αμερικανικό πρόγραμμα προστασίας. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ε, το κόστος των ζωοτροφών ποικίλει. Ως εκ τούτου αυτό θα πρέπει να συνυπολογίζεται στον τελικό ορισμό τιμής. Ελέγχθη επίσης ότι η αστάθεια των τιμών, μάλλον η διακύμανσή τους περισσότερο, είναι ένα εργαλείο που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει και εγώ διαρωτώ με ένα ευαίσθητο στοιχείο όπως είναι ο Γιώργος, μέχρι πού μπορεί να αντέξει τη διακύμανση των τιμών και πόσο χρειάζεται η διακύμανση των τιμών για να λειτουργεί η αγορά και για να μην προκύπτουν μετατοπίσεις τις οποίες έχουμε βιώσει κατά το παρελθόν στη γεωργική πολιτική και που σε τελική ανάλυση δεν οδήγησαν πουθενά όσον αφορά τις ε, χρηματοπιστωτικές αγορές. Το βρίσκω πολύ σημαντικό το ότι πρέπει στην Ευρώπη να σκεφτούμε ποια μπορεί να είναι η συνεισφορά των χρηματοπιστωτικών αγορών. Να σας θυμίσω όμως το παρελθόν είχαμε συζητήσεις ε, δυσάρεστες όπου ε, υπήρξαν πολλές ε, διατάξεις, θεσπίστηκαν διατάξεις και πολλοί πίστευαν και εδώ ότι το hedging η κάλυψη ε, είναι κάτι το δυσάρεστο, η κάλυψη κινδύνων ε, και ε, αντίστοιχη ήταν και η νομοθεσία που θεσπίστηκε. Έχω ένα ερώτημα γιατί δεν το κατάλαβα καλά. Ερώτημα προς τον Γενικό Γραμματέα. Μιλήσατε για αντικυκλικές πληρωμές. Εγώ δεν κατάλαβα ακριβώς τι εννοείται. Εννοείται ότι θα πρέπει να υπάρξει και πάλι συσχετισμός, δηλαδή αν ε, δεχόμαστε τις ανκυκλικές πληρωμές θα πρέπει να πιάσουμε κάθε ένα μεμονωμένο προϊόν να δούμε πού είναι υψηλή τιμή και πού είναι χαμηλή και η παρέμβαση να γίνεται όπου υψηλή η τιμή είναι χαμηλή ή μήπως εσείς με αντικυκλικές πληρωμές εννοούσατε παρέμβαση στο εισόδημα όταν πέφτει το εισόδημα. Κοιτάξτε, τα λέω αυτά από το πρίσμα του Γεωργού. Ε, δηλαδή θα μπορούσε κανείς να πει εξοικονομήσαμε 7 δις, ε, αλλά ε, αυτό ε, δεν θα σήμαινε απαραίτητα ότι εξοικονομήσαμε 7 δις. Δεν θα άρεσε στους γεωργούς. Δεν μπορώ ακριβώς ε, να καταλάβω ε, πού είναι το μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του συστήματος. Κυρία Ντελάε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με πρόλαβε ο κύριος Ντόρφμαν. Την ίδια ερώτηση είχα και εγώ. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε το θέμα της διαφάνειας δηλαδή σε ποιο επίπεδο και σε, ε, ποια φάση του κλάδου ε, έχουμε κάτι τέτοιο, γιατί στα οπορικεπευτικά, για παράδειγμα, κάθε φορά που προσπαθήσαμε να αποκαταστήσουμε διαφάνεια, ωφελούσαμε τις αλυσίδες διανομής. Εξηγήστε μας λοιπόν αυτό το θέμα της διαφάνειας. αναφέρθηκε το θέμα της αποταμίευσης, προληπτική αποταμίευση ή κάθε μορφή αποταμίευσης. Η φορολογία όμως δεν εμπίπτει στις κοινοτικές αρμοδιότητες, αλλά είναι αποκλειστική εθνική αρμοδιότητα. Οπότε τι μηχανισμούς θα μπορούσαμε να προβλέψουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δυσκολία. Γιατί κάθε κράτος, επαναλαμβάνω, έχει εθνική αρμοδιότητα για τη φορολογία. Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Ο κύριος Τεραμπέλα. Ευχαριστώ. Ε, με μένα τα πράγματα είναι απλά. Γιατί ερώτηση δεν έχω, αλλά θα εξαντλήσω τα δύο-τρία λεπτά για να σας εκφράσω τη δυσφορία μου. Γιατί μετά τις ε, παρουσιάσεις, τις έγκριτες παρουσιάσεις ε, των εμπειρογνωμόνων μας, Φερέρ, Φέντον, Αντινόλφι, Μπέισε, Καρλ, έγινε μια σωστή ανάλυση του φαινομένου, ε, αλλά λύσεις ε, λίγες ε, προτάθηκαν. Σχεδόν έχω πάθει κατάθλιψη γιατί εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας διαβεβαίωσε ότι είμαστε στο δρόμο, ότι αστάθηκαμε ανέκαθεν. Εννοείται, η αστάθεια των τιμών είναι γενής με τη γεωργία. Αλλά το θέμα είναι ότι αυξήθηκε υπερβολικά τα τελευταία χρόνια. Και η αστάθεια επιτόπου είναι από τους χειρότερους εχθρούς του γεωργού και κυρίως των νέων γεωργών ή ε, αυτών που εγκαταλείπουν τα χωράφια γιατί υπάρχει μία μόνιμη ε, αβεβαιότητα του γεωργικού εισοδήματος. Και δεν είναι κάτι καινούριο η αστάθεια στο γαλακτοκομικό τομέα. Εδώ και δύο ε, μήνες έχουμε τιμή στο γάλα που είναι κάτω του, του κόστου ε, και τη τιμή παραγωγή. Έχουμε ε, αγγίξει τον πάτο στο γάλα, έχουμε φτάσει στο αναδύρ. Οπότε κρίση υπάρχει και μάλιστα είναι βαθύτατη και α μα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είμαστε στον δρόμο και τα δίκτυα ασφαλείας δεν είναι αποτελεσματικά, δεν είναι ρεαλιστικά. Ρεαλιστές είναι οι Αμερικανοί. Άλλοι παγκόσμιοι εταίροι είναι πιο αποτελεσματικοί. Όλοι έχουν συνδέσει τις ενισχύσεις. Μόνο εμείς ε, σφυράμε κλέφτηκα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να μας πείσει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Και η πλειοψηφία των κυβερνήσεων ε, δεν θέλει να αλλάξει τίποτα. Είμαστε απομονωμένοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε την ΚΑΠ. Και θέλουμε μία θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που να είναι προοδευτική, να ανταποκρίνεται στην κρίση που βιώνει ο γεωργικός κόσμος ε, και μάλιστα ε, να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες των πραγματικών γεωργών, αυτών που βρίσκονται στα χωράφια, όχι των υπαλλήλων που δεν έχουν ε, δει στη ζωή τους και έχουν, βρίσκονται μόνο στα γραφεία και είναι άσχετοι με την πραγματικότητα. Δεν θέλω να προφέρω τη λέξη αυτιστικός, γιατί πραγματικά αυτό θα ήταν προσβολή για τους γονείς ε, των αυτιστικών παιδιών. Αλλά δεν μπορεί να συνεχίζει αυτή την πολιτική, αυτή τη στάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν προβλήματα στη Γεωργία, θα πρέπει να βρούμε λύσεις. Δεν ξέρω αν θα είναι οι αντικυκλικές ενισχύσεις, αν θα είναι τα ασφαλιστικά συστήματα. Θα τα αναλύσει φαντάζομαι όλα αυτά η κυρία Τελέ. Αλλά το μα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει και να προσπαθεί να δικαιολογήσει την παρούσα πολιτική. Αυτό πραγματικά είναι τελείως αλλοπρόσαλο και παλαβώ. άλλε ερωτήσει δεν έχω. Σα ευχαριστώ θερμά, αλλά πραγματικά δεν αξίζει να χώνεστε τόσο, κύριε Ταραμπέλα, και να εκνευρίζεστε. Ο κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα τους εμπειρογνώμονές μας ε, και υποβλήθησαν πολλές προτάσεις ε, για τα ασφαλιστικά συστήματα, για σύσταση ξεχωριστού ταμείου, για αποταμιεύσεις. Αυτά μπορεί να είναι καλά ως ε, θεωρητικό σημείο αφετηρίας. Επίσης αναφέρθηκε η ασφάλιση ε, ενός ποσοστού περιθωρίου κέρδους. Τι ποσοστό όμως εννοείται, 10%, 5%? περιθώρια, να ασφαλίζουμε. Επίσης ακούσαμε ότι τα ασφαλιστικά συστήματα θα πρέπει να ενεργοποιούνται ακόμη και όταν οι τιμές είναι υψηλές. Πάντως, για πολλά χρόνια τα γεωρικά εισοδήματα είναι τόσο χαμηλά και οι τιμές των γεωρικών προϊόντων τόσο χαμηλές, ώστε ο κόσμος ε, ε, έχει πρόβλημα και επιβίωση. Πώς μπορούμε να μιλάμε για αποταμίευση όταν δεν τα βγάζουν πέρα ούτε για το βιοπορισμό τους και τα ασφαλιστικά συστήματα πότε θα πρέπει να, ε, πότε θα πρέπει να ενεργοποιηθούν. Ε, θα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλία τα κράτη-μέλη ή να κάνουν τα κοινοτικά θεσμικά όργανα τις πρώτες ε, πληρωμές και να προσκαλέσουν τους γεωργούς ή να περιμένουμε μήπως να αυξηθούν, να ανέβουν οι τιμές. Στο μεταξύ όμως θα εξαφανιστούν ολόκληροι κλάδοι της γεωργίας ή της κτηνοτροφίας στα κράτη-μέλη αν περιμένουμε να αυξηθούν οι τιμές. Δεν κατάλαβα τη σύγκριση που κάνατε με τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ε, με το γαλακτοκομικό τομέα. Για μένα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Άλλο το ηλεκτρικό ρεύμα, άλλο ηλεκτρική ενέργεια και άλλο το γάλα. Άλλο γαλακτοκομικό τομέα. Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι μα πιέζει ο χρόνο. Και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα στοιχειώδε ε, γεωργικό εισόδημα για να μπορέσουν οι γεωργοί μα να επιβιώσουν. Και θα πρέπει να προσφέρουμε και μία λύση. Τι περιμένουμε, περιμένουμε να εξαρθρωθεί ολόκληρος ο κλάδος γεωργίας. Ε, θα πρέπει ε, να θρέφουμε τα ζώα μας. Δεν μπορούμε να τρέφουμε τις αγελάδες ε, μέρα παραμέρα με αφορά το μήνα. Τα ζώα χρειάζονται τροφή. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις καθημερινές ανάγκες και τα προβλήματα των γεωργών και κτηνοτρόφων. Ο κύριος Γιάρ. Κύριε Πρόεδρε, έχω κάτι να ρωτήσω που αφορά στη σταθερότητα των συστημάτων. Διότι ανεξάρτητα με το τι κάνουμε και πώς το κάνουμε, είτε πρόκειται για εξασφάλιση τιμών στο χρηματιστήριο, είτε με άλλους τρόπους εξασφάλιση, τα συστήματα πρέπει να είναι σταθερά. Γιατί δεν έχει κανένα νόημα ε, να εισάγουμε συστήματα τα οποία μετά από δύο-τρία χρόνια καταραίουν. Ένα λοιπόν πρόβλημα που ετέθη είναι το εξής. Ε, πώς μπορούμε μια υψηλή τιμή να τη διατηρήσουμε στην αγορά. Ε, ετέθη το θέμα των εξασφαλίσεων και βεβαίως ε, στην περίπτωση αυτή μπορεί κανείς να φανταστεί ένα σύστημα πολλών διαβαθμίσεων. Δηλαδή δεν θα πω απαραίτητα ένα σύστημα αστικής ευθύνης, όχι κάτι τέτοιο υπάρχει ας πούμε στη Γεωργία τη δυνατότητα ο ίδιος ο Γεωργός ε, να εξασφαλιστεί για τις αγελάδες του. Υπάρχει μια σχετική ασφάλεια. Ε, μπορεί να υπάρχει λοιπόν ένα μεικτό σύστημα αν θέλετε. Εγώ αυτό έχω να προτείνω. Και εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις. Το βασικό πρόβλημα ε, της σταθεροποίησης του εισοδήματος ε, είναι πώς θα το εξασφαλίσουμε χωρίς να παραβιάσουμε ε, τους ε, κανόνες της αγοράς και πώς θα εξασφαλίσουμε την επιστηστική ασφάλεια και εξορρόπηση προσφοράς και ζήτησης. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε δίκαιη φορολόγηση των εισοδημάτων των γεωργικών για να δώσουμε την ευκαιρία στους γεωργούς να εκπέσουν κάποιες ζημίες, να τις συνυπολογίσουν και θα πρέπει να βρούμε μηχανισμούς ε, για να εξασφαλίσουμε κάποια βεβαιότητα, κάποια σταθερότητα αντιμετωπίζοντας αυτές τις διακυμάνσεις. Ε, έχουμε κάποια συγκεκριμένη πραγματικότητα στις αγορές. Πώς θα αντέξουν οι γεωργοί αυτή την αστάθεια και αυτές τις, ε, διακυμάνσεις των τιμών. Είναι απαραίτητες για την λειτουργία της αγοράς. Ασχοληθήκαμε πολύ με τα χρηματοπιστωτικά και τα δημοσιονομικά μέσα. Ε, ίσως θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους δανειοδότησης, άλλες μορφές για να εξασφαλίσουμε αυτή τη σταθεροποίηση. Χωρίς όμως παρέμβαση στις γεωργικές αγορές δεν θα καταφέρουμε να λειτουργήσουμε. Και έδειξαν τα στοιχεία τα οικονομικά ότι δεν μπόρεσαν οι Γεωργοί μόνοι, τους να, μόνοι τους εξασφαλίσουν τη σταθερότητά τους. Χρειάζονται κάποιο είδος σε δημόσιες μέσω και του τραπεζικού, του δημοσιονομικού συστήματος. Βέβαια, ωραία ακούγεται να λέμε ότι θέλουμε ε, να κάνουμε μια σωστή εξασφάλιση για να αντιμετωπίσουμε τις ισχνές αγελάδες όταν έχουμε την εποχή των παχιών αγελάδων, αλλά αν έχουν και άλλη δουλειά οι δεν θα ασχολούνται οι ίδιοι με τη σταθεροποίηση του γεωργικού του εισοδήματο. Έχουν και άλλες ασχολίες. Επίσης, ε, σε ποιο βαθμό τα μέτρα αυτά θα είναι εθνικά ή ε, κοινοτικά, γιατί έχουμε κοινή γεωργική πολιτική, έχουμε ενιαία αγορά, οπότε η περισσότεροι από του μηχανισμού αυτού θα πρέπει να εφαρμόζονται σε κοινοτικό επίπεδο. Παρόλο που κάποιε ενέργειε θα πρέπει να γίνουν και σε εθνικό εννοείται. Αυτά και θα δώσω το λόγο και πάλι στον Διευθυντή τον κύριο Χανιώτη και κατόπιν στους εμπειρογνώμονε μας και πάλι με τη σειρά που μίλησαν και προηγουμένω Κύριε Χανιώτη, παρακαλώ έχετε το λόγο. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου ξαναδίνετε το λόγο. Ε, δεν θα σταθώ σε προσωπικά σχόλια και θα ρωτήσω μόνο το εξή. Αν θέλουμε να κάνουμε μια συζήτηση, ένα διάλογο για όσα συμβαίνουν στον πραγματικό κόσμο, θα πρέπει να βασιστούμε σε στοιχεία και γεγονότα. Αυτό ακριβώ προσπάθησα να κάνω και εγώ με τα όσα σα παρουσίασα. Που όλα μπορείτε να τα παληθεύσετε. Να υπενθυμίσω λοιπόν στον κύριο Ταραβέλα τα εξή. Όταν το 2008 όλοι έλεγαν ότι οι τιμές ε, της παγκόσμιας αγοράς, ε, τότε με τι παγκόσμιε τιμές αγοράς, ότι ο κόσμος δεν έχει πια φαγητό, ε, λέγαμε όχι δεν είναι θέμα της ζήτησης, είναι θέμα της προσφοράς. Εκεί να και το, η κρίση. Όταν όλοι έλεγαν ότι οι, γεωργοί δεν χρειάζονταν στήριξη των εισοδημάτων του, γιατί οι τιμές πόλη ήταν πολύ ψηλέ, τότε εμεί ήμασταν η πρώτη βάση του γραφήματος που είδατε, που λέγαμε γιατί έχουν επιδεινωθεί οι συνθήκε. Και αυτό ακριβώ σα είπα, συν 10% για τη γεωργία, συν 100% για τα λοιπάσματα και την ενέργεια. Όταν κανεί δεν έχει ακούσει καν για το Ελνίνιο, εμεί είχαμε κάνει υπόθεση για το για τον αντίκτυπο του Ελνίνιο. Όταν η Κίνα είχε 10% ανάπτυξη, εμείς ε, τρέχαμε το σημείο ότι 7% ανάπτυξη. Και όλα αυτά τα στοιχεία είναι διαθέσιμα, δημοσίως προσβάσιμα. Το ίδιο ισχύει και για την αστάθεια. Στη βιβλιογραφία λοιπόν εκεί έξω μπορείτε να βρείτε πολλές μελέτες που λένε ότι έχει αυξηθεί η αστάθεια και πολύ προσθέσω από ότι αυτές που λένε ότι ε, έχει μειωθεί η αστάθεια. Ό,τι και να λένε οι μελέτες όμως ένα είναι το, το σίγουρο το κατά πόσο μπορούμε να αξιολογήσουμε αν έχει δουλέψει και λειτουργήσει ε, μια πολιτική. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να εξετάσουμε τα στοιχεία. Για παράδειγμα, στις αμερικανικές πολιτικές το γαλακτοκομικό καθεστώς που αναφέρατε πολύ δείχνει ότι δεν λειτουργεί καλά και ότι δεν είναι δημοφιλές ανάμεσα στους αγιοργούς γιατί αφορά μόνο το ε, εθνικό επίπεδο και όχι το επίπεδο της εκμετάλλευσης. Αυτή τη συζήτηση να κάνουμε λοιπόν. Ενώ έχουμε δεύτερο, στο δεύτερο πυλώνα εργαλεία διαχείριση κινδύνου που αφορούν ακριβώ, αντιμετωπίζουν την αστάθεια εισοδημάτων για του γεωργού, δεν είναι δημοφιλή ούτε στη, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στη ΣΥΠΑ. Πολύ μικρό ποσοστό γεωργών το ακολουθούν. Ενώ ένα πολύ διαφορετικό σύνολο μέτρων πολιτική έχει ε, αποτελέσματα από πλευρά ε, διάρθρωση αγορά και από πλευρά εισοδημάτων των γεωργών. Και ο μόνο τρόπο, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, να κάνω αυτή τη συζήτηση είναι αν θέλουμε να συζητήσουμε δεδομένα και όχι απλώ να ανταλλάσσουμε κατηγορίε. Σα ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά. Οι εμπειρογνώμονε μα τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε συνεχίζω από την τελευταία φράση του κυρίου Χανιώτη που λέει ασχοληθούμε με τα στοιχεία, τα πραγματικά περιστατικά». Η αστάθεια που είδαμε σε πολλά προϊόντα και ήδη πρώτη ανάγκη στην Ευρώπη ξεκίνησε με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του 2003 στην Ευρώπη. Πριν το 2003 δεν είχαμε αστάθεια τιμών, είχαμε απλώς διακυμάνσεις. Σημείο και στοιχείο πρώτον. Πρόκειται για πολιτικό θέμα και τι πολιτική εφαρμόζουμε. Αυτή επηρεάζει την αστάθεια πραγματικά περιστατικά. Αν δεν κάνουμε τίποτα, έχουμε και θετικές και αρνητικές περιόδους. Και όταν φτάνουμε σε αρνητικές περιόδους, ε, έχουμε πάυση δραστηριοτήτων, έχουμε χρεοκοπίες γεωργών και γενικώ έχουμε μία αναδιάρθρωση, όπως το λέμε. Το πολιτικό ερώτημα είναι, θα δεχόμαστε σε κάθε κρίση αρνητικής αστάθειας μία αναδιάρθρωση των τρόπων παραγωγής ή των μέσων παραγωγής σε κάθε κράτος μέλος. Επίσης, ε, Καλό θα ήταν να αποφύγουμε αυτόν τον κίνδυνο. Γιατί πολιτικό δεν θέλουμε να βιώνουμε αναδιάρθρωση της παραγωγής κάθε φορά που έχουμε καταστροφική κρίση. Φυσικά θα πρέπει να τηρήσουμε τις ε, διεθνείς μας δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, τα διάφορα κουτιά του ΠΟΕ, το άνοιγμα των αγορών και ούτω καθεξής. Και γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε και κάποια μέσα. Όταν μιλούμε για τη φορολογία. Η φορολογία σήμερα ε, δεν ρυθμίζεται σε κοινοτικό επίπεδο, σε ενωσιακό επίπεδο, αλλά σε εθνικό. Είναι θέμα πολιτική απόφαση. Εμεί είμαστε απλοί εμπειρογνώμονε. Τι να σα πούμε, δεν έχουμε εμεί δικαίωμα να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει και με τι ασφάλειε. Επαφίονται στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών. Οι ασφαλίσει. Επίση, η φορολογία σίγουρα θα, είναι, θα ήταν ένα εξαιρετικό μέσο για να επανισορροπήσουμε τα πράγματα και ε, να εξασφαλίσουμε μια βιωσιμότητα των ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων απέναντι στις ε, σοβαρές διακοιμάνσεις και στην αστάθεια. Και όταν μιλούμε για εξασφάλιση του περιθωρίου κέρδους, δεν μιλούμε για θεωρητικό περιθώριο, αλλά για το πραγματικό, το ιστορικό περιθώριο κέρδους κάθε εκμετάλλευσης. Και η ασφάλεια που θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη και να καλυφθεί από δημόσια κονδύλια όπως συμβαίνει σε μερικές χώρες, αφορά αφενός ε, την κάλυψη ενός ποστού 65% ε, του, των, ε, των χρεολυσίων που καταβάλουν οι γεωργοί και επίσης σε περίπτωση σοβαρών κρίσεων θέσπιση δημόσιας αντασφάλισης ώστε να μην μετακυλίουν το κόστος της ασφάλισης οι αντασφαλιστές στους ασφαλισμένους. Το θέμα λοιπόν είναι τι πολιτική θέλετε να θεσπιστεί και να εφαρμοστεί. Και γι' αυτό είστε αρμόδιες ίσως πολιτικοί να, να απαντήσετε και όχι εμείς οι εμπειρογνώμονες. Ευχαριστώ κύριο Σαντινόλφη. Ε, ε, Κοιτάξτε, θα ήθελα να πω το εξής. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη ως πολίτη. Το θέμα της εξοικείωσης, αυτό που παρουσιάζουμε τύρα, ε, κατ' ουσίαν είναι, σημαίνει ότι προσπαθούμε να παρουσιάσουμε λύσεις αλλά και προκλήσεις όπως αυτό που έχει σχέση με το ε, σύστημα που χρησιμοποιείται για την ηλεκτρική ενέργεια. Πολλές φορές ε, τα συστήματα που παρουσιάζονται κρύβουν πάρα πολλά. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να πω. Και το δεύτερο είναι ότι κατά την άποψή μου εδώ υπάρχει και κάποια νοσταλγία ε, σας λέω ότι είναι μια προσωπική μου άποψη αυτή, δηλαδή κινδυνεύουμε να είμαστε μη δημοφιλείς, ε, κυρίως ε, σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος ε, Χανιώτης, γιατί κατά την άποψή μου υπάρχει κάτι σημαντικό. Αυτές οι μικρές ε, καινοτομίες που έχουν προκύψει έχουν σχέση με το stabilization tool και επίσης και με μια εργαλειοθήκη για την σταθεροποίηση. Το να ψάχνουμε να βρούμε μια λύση αυτό δεν είναι λάθος, γιατί το να ψάχνουμε να βρούμε τόσο ισχυρούς μηχανισμούς σταθεροποίησης όπως συνέβη ε, κατά το παρελθόν, αυτό σας λέω πραγματικά είναι τρέλα και αυτό νομίζω μπορώ να το πω ως άποψή μου. Να διευκρινίσω κάποιες από τις αναφορές για την ε, αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Να ξεκαθαρίσω. Στα περισσότερα γεωργικά προϊόντα ακολουθούμε την οριακή ε, τιμή κόστους αν υπάρχει υπερβολική παραγωγή, τότε η τελευταία μονάδα προσφοράς είναι που ορίζει την ε, αγορά. Γιατί δεν θέλουμε να υπάρξει κατάχρηση. Σε αρκετέ περιπτώσει ήθελαν να συμμετάσχουν ε, συνεταιρισμοί και η Επιτροπή είπε όχι, είναι επικίνδυνο. Στην αγορά ηλεκτρική ενέργεια δίνουμε δυνατότητα στην ρυθμιστική αρχή να κάνει τη μέση τιμή, να την καθορίσει και για αυτό το είδος, ε, για αυτό το τμήμα του, της τιμής κόστους, ε, το πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας δεν βασίζεται στο κόστος του πλεονάσματος εκείνη τη στιγμή. Πρόκειται για τιμολόγηση ισχύω. Και πολλές φορές άκουσα τη σχέση για αυτό με το γεωργικό τομέα. Για ορισμένα προϊόντα, ε, ιδίω τα, τα, πολύ αναλώσιμα, στα απορροκυπευτικά, επιτρέπουμε και στι οργανώσει παραγωγών να κάνουν αυτή τη μεσοστάθμιση τη κοστολόγηση για τα επιχειρησιακά του προγράμματα για να αποσύρουν προϊόντα από την αγορά. Επομένω υπάρχει διαφορά όντω. Στην ηλεκτρική ανάργεια ε, έχουμε την... Η μονάδα μέτρηση είναι τα λεπτά, ενώ στα γεωργικά είναι ε, τα χρόνια. Αλλά πέραν τούτου, άμα το εξετάσουμε ευρύτερα, πρέπει να τα συγκρίνουμε τα δύο συστήματα. Δεν είναι τα ίδια, αλλά μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Ένα από τα θέματα είναι ότι στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και στα αγορικευτικά, επειδή θέλουμε συνεχή προσφορά, επιτρέπουμε σε ένα βαθμό την ε, μεσοστάθμιση της κοστολόγησης, το οποίο δεν επιτρέπουμε για πολλά ε, οπορικευτικά. Δεν λέω ότι αυτό θα πρέπει να γίνει για όλα, όμως μπορούμε τουλάχιστον να το εξετάσουμε. Um, I think Mr. Dorfman uh, raised Νομίζω ότι ήταν πολύ εύστοχο το σχόλιο του κ. Ντόρφμαν για την πληθώρα των κανονισμών που πλαισιώνουν τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Ε, και εμείς ε, ε, ως εμπορική επιχείρηση υφιστάμεθα την ίδια ρύθμιση με τις τράπεζες, τις μεγάλες τράπεζες και δεν έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε. Γιατί πρόκειται για μερικές εμπορικές εταιρείε που μικρής εμβέλειας που έχουν υποχρεώσεις να τηρούν κανονιστικές ρυθμίσεις που ισχύουν για μεγάλες τράπεζες. Επίσης, πώς μπορεί ένα συνεταιρισμό να εγγυηθεί μια τιμή 36 λεπτά το λίτρο το γάλα για τον Γιώργο. Δεν είναι ο συνεταιρισμό που αναλαμβάνει το κίνδυνο. Ο συνεταιρισμό διευκολύνει την πρόσβαση του Γιώργου στην αγορά. Γιατί όπως και οι χώρες όπου έχουμε με έναν γεωργό, με έναν κτηνοτρόφο με 15 ε, αγελάδες, να έχει την ίδια πρόσβαση με αυτόν που έχει κοπάδι με χιλιάδες ε, αγελάδες ζωικό κεφάλαιο, να έχει την πρόσβαση αυτή και ο μικρός κτηνοτρόφος μέσω του συνεταιρισμού. Βέβαια, τον κίνδυνο δεν τον φέρει ο συνεταιρισμός, αλλά μετακυλεί τον κίνδυνο στην αγορά ο συνεταιρισμός. Εγώ αναφέρθηκα στα πλεονεκτήματα των χρηματοπιστωτικών ε, μέσων. Βέβαια δεν είναι πανάκια, δεν είναι θαυματουργή λύση, ούτε είναι εύκολο να εφαρμοστούν, αλλά μπορούν να αποτελέσουν τμήμα της λύσης. Οι υπόλοιπε λύσεις αφορούν τις ασφάλειες και άλλα μέτρα. Και αυτά τα μέτρα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για να εξασφαλιστεί πρόσβαση του Γεωργού σε διάφορους τρόπους ε, ε, διαχείρισης της κρίσης, της αστάθειας των Δημών. Δεν υπάρχει μία μόνο λύση θαυματουργή. Και σίγουρα θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια ανταγωνιστικότητα μεταξύ των λύσεων, ώστε να κάνει επιλογή κόστου-οφέλου και ο Γεωργό και η Ευρωπαϊκή Ένωση των διαφορών μέσων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι ΗΠΑ και τη Νέα Ζηλανδία, χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία και ανταγωνίζονται στην ίδια αγορά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο και η Κίνα και άλλε χώρε θέλουν τέτοια μέσα για να εξυπηρετήσουν και τους καταναλωτές. Οπότε αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων και να αντιμετωπίσουμε την αστάθεια των τιμών θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και στο δικό μας κλάδο την πρόσβαση σε τέτοιου είδους χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Ευχαριστώ. Μάλιστα, άκουσα τα όσα ανέφερε ο κύριος Χανιώτης ε, πολύ λογικά τα όσα αναφέρει, αλλά δυστυχώ δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, το οποίο επεσήμανε και ο κύριο Ταραμπέλα και ο κύριο Φερέρ. Εδώ υπάρχει μια κατάσταση συνεχού ε, κρίση. Αυτό είναι το πρώτο. Όταν συγκρίνουμε μέσα, όταν ε, συγκρίνουμε την, τα γεωργικά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια, υπάρχουν πολλά στοιχεία ισοδυναμίας. Είναι δύσκολο βέβαια να συγκρίνουμε τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όπου έχουμε μερικούς μόνο εμπορευομένους και στον γεωργικό κλάδο που έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες παραγωγούς. Πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου. Μετά υπάρχει ε, μία επιλογή το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να επιλέξουν μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη Γεωργία. Δεν έχουμε στρατηγική, έχουμε μηχανισμούς παρέμβασης μόνο, όχι στρατηγική. Και αυτό είναι κρίμα, ενώ όλε οι υπόλοιπε μεγάλες χώρες έχουν στρατηγική. Αν δείτε την εξέλιξη της δημόσιας ε, κοινή γνώμης ε, για τη γεωργία σε υπόλοιπες χώρες, είναι μεγάλη αύξηση γιατί είναι ε, πολύ σημαντικό στρατηγικός κλάδος και σε, μια, σε έναν κόσμο με δέκα δις ε, πληθυσμό δεν γίνεται να μην το προλέψουμε αυτό. Πρέπει να γίνει μια πολιτική και στρατηγική επιλογή. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το ρυθμίζουμε τα πάντα όπως το παρελθόν. Πρέπει να τα ρυθμίζουμε με διαφορετικό τρόπο. Και αυτό γίνεται με ε, αντίστοιχου ή και χαμηλότερου προπολογισμού. Πρέπει να γίνει. Αυτό είναι απολύτω παρέτο. Και για να απαντήσω στον κύριο Ντόρφμαν, έδωσα στην ε, Γενική Γραμματεία τη Κομισιόν συγκεκριμένα έγγραφα που αντιμετωπίζουν τον αφορούν τον αντίκτυπο των όσων κάνουμε στα δημητριακά, στα γαλακτοκομικά και σε άλλους κλάδους. Για την περίοδο 2011-2015 οι ε, επιπτώσεις ήταν 10 ε, δις κάθε χρόνο και βλέπουμε ότι θα διατηρούσαμε τα μέσα ε, εισοδήματα σε ένα σταθερό επίπεδο για τα επόμενα πέντε χρόνια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους γεωργούς. Κάτι τελευταίο. Αστάθεια τιμών ή εισοδημάτων. Βεβαίως αν υπάρχει μεγάλη στάθεια των τιμών αυτό θα επηρεάσει και τα εισοδήματα. Γιατί αφού και οι ενισχύσει είναι αποσυνδεμένε από τι τιμέ, είναι πάντα σχεδόν οι ίδιε. Η μόνη εξέλιξη είναι η εξέλιξη ω προ τη σύγκληση σε συγκεκριμένα κρατημέλη. Επομένω, η επίπτωση των τιμών στα εισοδήματα είναι άμεση. Όταν οι τιμές είναι πολύ ε, χαμηλές, δεν φτάνουν ε, οι ε, και όταν είναι πολύ ψηλές επίσης δεν έχουν τα, τις απαραίτητες επιπτώσεις και αντίκτυπο το Κοινοβούλιο, η Κομισιόν και το Συμβούλιο θα πρέπει να τα προσδιορίσουν όλα αυτά στο μέλλον. Θα υπάρχει μια σύνδεση για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλά σε σχέση με τον ε, ΠΟΕ βλέπουμε ότι είναι απόλυτα συμβατό με τον ΠΟΕ, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αξιοποιεί ε, την ε, ρήτρα ντεμίνιμης που ακολουθείται στον ΠΟΕ. Ευχαριστώ. <coughs> Νομίζω ότι ε, τώρα άναψη συζήτηση και δυστυχώς ο χρόνος μας τελειώνει. Και σίγουρα δεν υπάρχει απόλυτη σύμπνοια, υπάρχει αρκετή διάσταση απόψεων. Γι' αυτό εκείνο το ερώτημα. Έχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο έναν τρόπο διαχείρισης α, της αστάθειας των τιμών, αλλά είναι τελείως διαφορετικές οι προκλήσεις. Έχουμε διάφορα επίπεδα. Έχουμε το κοινοτικό, το εθνικό και το τοπικό. Και τα τρόφιμα ακολουθούν ε, την ε, πορεία των αγορών, γιατί τα τρόφιμα είναι υλικά προϊόντα, δεν είναι άειλα προϊόντα όπως είναι τα χρηματοπιστωτικά. Οπότε δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα τρόφιμα με τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Επίσης, τι ε, πορεία πρέπει να ακολουθήσει η κοινή γεωρική πολιτική ώστε να εξασφαλίσει και τη σταθεροποίηση ε, του εισοδήματο. Όχι σταθεροποίηση τιμών, αλλά σταθεροποίηση γεωργικού εισοδήματο. Ε, γιατί έτσι θα εξασφαλίσουμε και την επιστημιστική ασφάλεια. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, επιστημιστική ασφάλεια. Α μην το ξεχνούμε. Γιατί η κοινή γεωργική πολιτική έχει θετικά αποτελέσματα. Και Μερικές φορές βέβαια έχουμε κάποιες κρίσεις και θα πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε για να αφυπνιστούμε και να δούμε τα πράγματα με νέο πνεύμα. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ε, καλό κλίμα για την κοινή γεωρική πολιτική. Και το παράδειγμα είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός, οι τελευταίες δημοσιονομικές προοπτικές. 45 εκατομμύρια λιγότερα είχαμε. 11-12% μικρότερο προϋπολογισμό σε σχέση με το 2011. Ενώ ταυτόχρονα έχουμε μια διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, το θέμα του γεωργικού εισοδήματος είναι σημαντικό ή το μερίδιο των νέων γεωργών ε, στην αγορά. Πώς θα εξασφαλίσουμε παρουσία του στην αγορά αν δεν σταθεροποιήσουμε το γεωργικό εισόδημα θα μειώνεται ο αριθμός των νέων γεωργών, των νέων εισόδων. Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ανάλυση και ευχαριστώ τους εμπειρογνωμονές μας που ε, μας διαφώτισαν σε πολλά σημεία και θα τα αξιοποιήσουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ λοιπόν θερμά τους εμπειρογνωμόνες. Μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα, αλλά γι' αυτό γίνεται συζήτηση. καλό είναι με τη διάσταση απόψε να φωτίζονται διαφορετικές πτυχές ε, του θέματος στη συζήτηση. Είναι πολύ χρήσιμο κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα τα αξιοποιήσει η συγκεκριά μας, η κυρία Ντελαέ, κατά την εκπόνηση της έκθεσής της. Και, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να επιβεβαιώσουμε τώρα τα συμπεράσματα και τις αποφάσεις των συντονιστών που συνεδρίασαν πριν το μεσημέρι Σα στείλαμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα, τις αποφάσεις των συντονιστών. Ελπίζω να τις εγκρίνουμε. Αν δεν υποβληθούν αντιρρήσεις, ε, θα θεωρηθούν ότι εγκρίνονται οι αποφάσεις των συντονιστών. Διάφορα δεν υπάρχουν. Να υπενθυμίσω πότε θα γίνει η επόμενη μας συνεδρίαση, 14 και 15 Μαρτίου. 14 Μαρτίου 3 με 6.30 Επίσης, ε, μετά τις 5 θα γίνει η ψηφοφορία όπως μας ζήτησε ο κύριος ε, Νίκολσον και έχουμε και ολοήμερη συνεδρία στις 15 Μαρτίου. Ευχαριστώ θερμά τους εμπειρογνώμονες, σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή. Λύεται η συνεδρίαση, ευχαριστώ και τους δημιουργούς συνεπρόεδρους, ευχαριστούμε και εμείς. Καλό σας απόγευμα.